Καλησπέρα σε όλους. Ζητώ συγγνώμη που ξεκινούμε νωρίς τη συνεδρίασή μας, αλλά καμιά φορά υπάρχει μόνο μια δυνατότητα για να καταφέρουμε όλοι να μπορούν να συμμετάσχουν στις εργασίες μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκείνους από εσά που είναι παρόντες και είμαι σίγουρη ότι αργότερα θα καταφτάσουν και άλλοι. Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι απλώς η έγκριση της ημερήσιας διάταξης που θεωρώ ότι την υποστηρίζετε, δεν υπάρχει αντίρρηση. Δεύτερο θέμα είναι η έγκριση των πρακτικών της 19ης Οκτωβρίου του 2009. Δεν μας εκκοινοποιήθη κάτι, οπότε θεωρώ ότι εγκρίνονται και τα πρακτικά. Τρίτο σημείο είναι ανακοινώσεις της Προέδρου. Δεν έχω τίποτα να ανακοινώσω, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε. Πάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης και χαίρομαι που μπορώ να καλωσορίσω τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον Jean-Claude Trichet, για τη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων για τον νομισματικό διάλογο υπό την δική μου προεδρία. Οπότε, χωρίς να χρονοτριβήσω, θα δώσω το λόγο στον Jean-Claude. Ευχαριστώ, λέει ο κ. Τρισέ. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Νομισματικών και Οικονομικών Υποθέσεων, αυτή είναι η πρώτη συνάντησή μας μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Η νέα συνθήκη σίγουρα είναι ένας λόγος για να γιορτάζουμε στην Ευρώπη εν γέννη και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα κάνει την Ένωση ισχυρότερη, αποτελεσματικότερη, με καλύτερες επιδόσεις. Οι εξουσίες και ευθύνε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυξάνονται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επίσημα γίνεται θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και όλα τα βασικά της χαρακτηριστικά, πάνω απ' όλα η ανεξαρτησία της, είναι κάτι που επιβεβαιώνονται. Τώρα στα πλαίσια της ε, νέας συνθήκης χαιρόμαστε για τη συνεργασία μας τη μελλοντική με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ποιότητα αυτής της συνεργασίας ήταν υποδειγματική κατά την άποψή μου κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Λοιπόν, όσον αφορά θα ήθελα να πω κατά τα λοιπά ότι η αξιολόγησή μας όσον αφορά την οικονομική κατάσταση που ισχύει τώρα είναι κάτι που θέλουμε να εξετάσουμε. Δεύτερον, η στρατηγική μας εξόδου από την κρίση με την εκπνοή των νομισματικών μέτρων των εκτάκτων που ελήφθησαν και που έχουν εισαχθεί και εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της ακμής της κρίσης, είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε, και τρίτον, η συστημική κίνδυνη του όλου χρηματοπιστωτικού οικοδομήματος, του συστήματος. Θα ήθελα τώρα να στραφώ στις οικονομικές και νομισματικές εξέλιξεις. Η οικονομική κατάσταση και οι προοπτικές εξακολουθούν να βελτιώνονται μετά από την προηγούμενη ακροασή μας που ήρθα, όταν ήρθα εδώ σε αυτήν την Επιτροπή 10 η Ευρωζώνη ε, δείχνει όλο και περισσότερα σημεία ανάκαμψης. Η οικονομική δραστηριότητα το τρίτο ε, τρίμηνο θεωρείται ότι αυξήθηκε κατά 0,4% εν συγκρίση με το προηγούμενο τρίμηνο το 2010 αναμένεται να δούμε μια μέτρια ανάκαμψη. Αυτό ταιριάζει με, τα, με τις πρόσφατες προβλέψεις στο Eurosystem ε, που δημοσιεύτηκαν την περασμένη Πέμπτη. Όμως αυτές οι προσδοκίες περιβάλλονται ακόμα από πάρα πολύ αβεβαιότητα. Εν ώψη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα, οι κίνδυνοι για τις προπτικές και τις προβολές είναι γενικά ισορροπημένοι όσον αφορά τις εξελίξεις για τις τιμές, τον πληθωρισμό και τις πληθωριστικές πιέσεις. Αυτά παρέμειναν χαμηλά κατά τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τις προσδοκίες μας, ο πληθωρισμός ε, ξανά έγινε θετικός τον Νοέμβριο και φτάσαμε 0,6% ε, προσβλέπουμε να παραμείνει μέτριος ο πληθωρισμός όσον αφορά τον ορίζοντα που καλύπτεται τις πολιτικές μας σε συνδυασμό με την αρκετά χαμηλή ανάκαμψη της ζήτησης. Οι δείκτες των προσδοκιών πληθωρισμού μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ε, παραμένουν ε, σταθερές σύμφωνα με το στόχο του Διοικητικού Συμβουλίου να παραμείνει ο πληθωρισμός κάτω αλλά κοντά στο 2% μεσοπρόθεσμα. Η νομισματική μας ανάλυση επιβεβαιώνει την αξιολόγηση των χαμηλών πληθωριστικών πιέσεων μεσοπρόθεσμα. Και βλέπουμε ότι οι πιστώσεις και τα, η αύξηση των πιστώσεων εξακολουθεί να μειώνεται. Όσον αφορά τα στοιχεία που έχουμε, προβλέπουμε περισσότερη επιβεβαίωση ότι θα έχουμε χαμηλότερα επίπεδα ανάκαμψης. Και η αύξηση των δανείων προς επιχειρήσεις βλέπουμε ότι μένει πίσω από τον επιχειρηματικό κύκλο και έχουμε χαμηλά επίπεδα παραγωγής και αυτά μαζί με τη μεγαλύτερη βεβαιότητα όσον αφορά τις προοπτικές των επιχειρήσεων θα μειώσουν τη ζήτηση από πλευρά εταιριών για χρηματοδότηση από τράπεζε τον επόμενο μήνα, του επόμενου μήνε, κυρίω για βραχυπρόθεσμα δάνεια. Ε, ταυτόχρονα, η γενική χρηματοδότηση και οι συνθήκη χρηματοδότηση εξακολουθούν να βελτιώνονται και αυτό θα πρέπει να υποστηρίξει τη ζήτηση για δάνεια κατά την επόμενη περίοδο. Έτσι, επί του παρόντο δεν βλέπω να υπάρχουν σημάδια ε, πιέσεω μεγάλων προβλημάτων τη πιστώση στην Ευρωζώνη. Ε, παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ όμω όλε τι εξελίξει. Έχουμε αυτό το ιστορικό, το υπόβαθρο και το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να εξετάζει τι γίνεται με τα βασικά επιτόκια τη ε, Ευρωπαϊκή Σχετική Τράπεζα και κάνουμε τα δέοντα. Όσον αφορά την χρηματοσυντητική κρίση, όπως γνωρίζει η Επιτροπή, το Eurosystem έχει εισαγάγει διάφορα έκτακτα μέτρα από τον Οκτώβριο του 2008 και όπως σας εξήγησα προηγουμένως, τα πέντε βασικά στοιχεία της υψημένης υποστήριξης για τις πιστώσεις είναι ε, σταθερά επιτόκια, επέκταση του καταλόγου για και επίσης περισσότερα μέτρα για τη χρηματοδότηση, προβλέψεις για ρευστό σε ξένα νομίσματα και υποστήριξη μοτοστοτικών αγορών μέσω Μετρημένη αλλά σημαντικής, ε, σημαντικού προγράμματο για δημόσιες αγορές. Αυτά τα μέτρα εξυπηρέτησαν καλά ε, την οικονομία σε κρίσιμες στιγμές, ε, υποστήριξαν τη δυνατότητα των τραπεζών να παρέχουν πιστώσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης, εξασφαλίζοντας ότι οι χρήματα και οι συνθήκες για την αγορά τη χρηματοπιστωτική ταιριάζει με τα νομισματικά μέτρα και την πολιτική τη σχετική που αφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο. Γνωρίζετε τώρα τα έκτακτα μέτρα είχαν σαν στόχο να ε, ε, εκπνεύσουν σταδιακά και τώρα γίνεται με φυσικό τρόπο αυτή η εκπνοή και η λήξη των μέτρων και το παρόν πλαίσιο μα είναι αρκετά ευέλικτο, ώστε να είμαστε σε θέση να προσαρμοζόμαστε όσον αφορά τι συνθήκε ρευστότητα όταν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Η θεσμική μα ανεξαρτησία σημαίνει ότι είμαστε περιόριστοι όσον αφορά τη δυνατότητά μα να εφαρμόζουμε τα δέοντα μέτρα και αποφάσει. Πάντα τόνιζα ότι η σταδιακή εξάλληψη των μέτρων θα γίνει έγκαιρα και σταδιακά θα πρέπει να είναι έγκαιρη, διότι κάποιο δεν θα πρέπει να το κάνει αυτό πολύ νωρί, ούτε πολύ αργά. Ο, εκ των υστέρων εφαρμογή των μέτρων δεν, δεν είναι κάτι Σταδιακά πρέπει να γίνεται εξάλληψη των μέτρων διότι και η κατάσταση ε, βελτιώνεται σταδιακά. Την περασμένη Πέμπτη πήραμε μια απόφαση να ξεκινήσουμε σταδιακή πάυση κάποιων από, τον έκτακτον, από τα έκτακτα μέτρα ρευστότητα, διότι δεν χρειάζονται στον ίδιο βαθμό αυτά τα μέτρα όπω κατά το παρελθόν. Έτσι θα αποφύγουμε στρεβλώσει που συνδέονται με τη διατήρηση εκτάκτων μέτρων για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι σημαντικό λοιπόν να αποφύγουμε την κατάσταση κατά την οποία οι τράπεζες εξαρτώνται πάρα πολύ από έκτακτη χρηματοδότηση τη κεντρική τράπεζα. Στα πλαίσια λοιπόν τη σταθεροποίηση των νομισματικών αγορών και πρέπει να ενισχύσουμε τα κίνητα για τι τράπεζε να αναδιαθρώσουν τα ισοζύγια του, ούτω ώστε να γίνει ανακεφαλοποίηση. Πέραν αυτό, έγκαιρη και σταδιακή κατάργηση των μέτρων θα πρέπει να βοηθήσει τη δραστηριότητα στον νομισματικό τομέα και θα πρέπει να ενισχύσει τον έλεγχο, τον ισότιμο μεταξύ των διαφόρων τραπεζών. Αυτό είναι το όλο ιστορικό και γι' αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προσαρμόσει τον ε, σχεδιασμό κάποιων επιχειρήσεών μας αναχρηματοδοτήσεως. Θα συνεχίσουμε πλήρως να καλύπτουμε τις ανάγκες ρευστότητας των τραπεζών και να καθορίσουμε τα επιτόκια σε όλες τις επιχειρήσεις μας χρηματοδοτήσεως όσον αυτό είναι αναγκαίο και τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Απριλίου του επόμενου έτους. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε να παρέχουμε υποστήριξη ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ούτως ώστε να ευκολύνουμε την παροχή πιστώσεων στην Ευρωζώνη και στην οικονομία τη Όσον αφορά τι επιχειρήσει μα του ενό έτου, αποφασίσαμε να μην προβούμε σε περαιτέρω τέτοιε πέρα από αυτή του Δεκεμβρίου που ήδη ανακοινώθη. Οι βελτιωμένες συνθήκες όσον αφορά τι χρηματοστικές αγορές ε, δείχνουν ότι όλα δεν απαιτούνται στον ίδιο βαθμό τα μέτρα ρευστότητα όπως κατά το παρελθόν. Παρομοίως προτιθέμεθα να σταματήσουμε τι επιχειρήσει εξάμεινε αναχρηματοδοτήσεω μετά την τελευταία αυτή επιχειρήση που θα γίνει το τέλο Μαρτίου του επόμενου έτου. Επιτρέψτε μου να πω μερικά λόγια όσον αφορά τι ευρύτερε συνέπειε των αποφάσεων που έχουμε λάβει, όσον αφορά τα έκτακτα μέτρα, ε, εστιαζόμενος ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που είναι εκτός Ευρωζώνης, μακροοικονομικές και οικονομικές συνθήκες σε αυτές τις χώρες ε, φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί ε, παρόλο που υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην περιοχή αυτή. Ε, εν γέννη έχουν σταματήσει κεφαλοικές, δεν, μάλλον δεν σταμάτησε κεφαλοικές ροές προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη και η παρουσία ξένων τραπεζών έπαιξε σταθεροποιητικό ρόλο. Διότι σε μεγάλο βαθμό αυτές οι τράπεζες μπόρεσαν να κρατήσουν ε, την έκθεση του, την παρουσία του στην περιοχή. Η εκτετική και ε, τα μέτρα που δώσαμε όσον αφορά τη ευστοποίηση στην Ευρωζώνη συνέβαλε σε αυτή τη σταθεροποίηση. Και πέραν αυτού, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρήχε υποστήριξη ρευστότητα σε κάποιε κεντρικέ τράπεζε μη Ευρωζώνη σε περίπτωση τη λειτουργία των αγορών για να διευκολύνουμε ή για να διευκολύνουμε τη λειτουργία του διεθνούς Χρηματοδοτικού συστήματος. Τέλος, ε, θα ήθελα να προσθέσω και κάποια σχόλια όσον αφορά τις φορολογικές στρατηγικές διεξόδου. Πολλές κυβερνήσεις της Ευρωζώνης αντιμετωπίζουν υψηλές φορολογικές ανισορροπίες που αυξάνονται πάρα πολύ γρήγορα που δεν μπορούν να κρατήσουν μακροπρόθεσμα διότι μπορεί να μειωθεί η εμπιστοσύνη του κοινού όσον αφορά τη βεσιμότητα των δημοσιονομικών με αρνητικέ συνέπειε για το συνέστημα που κρατεί στην αγορά και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσχερέστερε μέσω, βραχυ... Ε, μακροπρόθεσμα επιτόκια και βιώσιμες, μη βιώσιμες φορολογικές τοποθετήσει, ίσω δυσκολέψει την νομισματική μα πολιτική για τη σταθερότητα των τιμών. Χρειάζεται αξιόπιστη στρατηγική φορολογική εξόδου από την κρίση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ούτω ώστε να υπάρχουν σωστά εδρεωμένε προσδοκίε. Τέτοιε στρατηγικέ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν αξιόπιστα μέτρα, κυρίω όσον αφορά τι δαπάνε. Και όσοι ενεφωνήθη από το Συμβούλιο Κοφίν την περασμένη εβδομάδα, οι κυβερνήσει θα πρέπει να καθορίσουν συγκεκριμένα ποσοτικέ ε, ποσοτικά μέτρα μάλλον, ποσοτικοποιημένα μέτρα για να γίνει βιώσιμη διόρθωση φορολογικών ανισορροπιών. Αρκετές χώρες θα πρέπει να συνεχίσουν το 2010 τις προσπάθειες για σταθεροποίηση και όλες οι άλλες το 2011 ε, το αργότερο για την ενοποίηση αυτών των μέτρων. Θα ήθελα κυρία Πρόεδρε να στραφώ προς το τελευταίο θέμα το οποίο επιλέξαμε, δηλαδή το θέμα του συστημικού κινδύνου σε χρηματοστικά συστήματα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Ο συστημικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνο ευρεία κατάρρευση του οικονομικού συστήματος και είναι αποτέλεσμα ε, παρεμπόδιση λειτουργίας του χρηματοστικού συστήματος που απορρέει από τον υψηλό βαθμό διασύνδεση και αλληλεξάρτηση μεταξύ των στοιχείων του συστήματος. Συστημικός κίνδυνος είναι κάτι διαφορετικό από τον κίνδυνο που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια και τη σωστή λειτουργία των μεμονωμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ε, περαιτέρω, συστημικός κίνδυνος όταν ε, παρουσιαστεί επηρεάζει σοβαρά τη, δια... τη δημοσιονομική διαμεσολάβηση, τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση σε τέτοιο βαθμό που υπάρχουν αρνητικές συνέπειες που ξεχυλίζουν και επηρεάζουν την πραγματική οικονομία έδειξε η κρίση ότι στομικός κίνδυνος ίσως να ξεκινά από τη συλλογική συμπεριφορά των διαφόρων θεσμικών φορέων και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική αγορά. Έχει δείξει τη σημασία που έχει η βελτίωση της γνώσης μας και της αξιολόγησης του, της διασύνδεσης των διαφόρων χρηματοπιστωτικών συστημάτων και μέσω άμεση σχέση μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και έμεση σχέσης που δημιουργείται στις σηματοπιστωτικές αγορές. Λοιπόν, η βασική αξιολόγησή μας που γίνεται κατά θεσμικό ίδρυμα έρευνα τη διαθεσιμότητα του κάθε φορέα σε διάφορα σενάρια ασκήσεως πιέσεων από αυτόν. Αντίθετα, η αξιολόγηση συστημικού κινδύνου έρευνα τη δυνατότητα όλο το σύστημα γενικά ή σημαντικά κομμάτια του συστήματος να είναι βάλωτα και θεωρεί ότι σημαντικός κίνδυνος μπορεί να προκύψει και από το ίδιο το χρηματοδοτικό σύστημα. Τέτοιοι κίνδυνοι μπορούν να προκύψουν, παραδείγματο χάρη, διότι μεγάλα κομμάτια του συστήματο ίσω να έχουν παρόμοιε εκθέσει. Μπορεί να βασίζονται στι ίδιε πηγέ χρηματοδοτήσεω, μπορεί να εκτίθενται σε αύξηση χρηματοπιστωτικών ανισορροπιών και μπορεί να συμπεριλαμβάνει πολλέ διαφορέ μεταξύ νομισμάτων και αξιογράφων που αυξάνουν το ευάλωτον του τομέα και μπορεί να εκτίθεται και σε υποαξιολόγηση, υποτίμηση και κακή τιμολόγηση και αξιολόγηση των κινδύνων. Η αξιολόγηση των συστημικών κινδύνων του χρηματοδοτικού συστήματος, δηλαδή πόσο στέρεα είναι η ίδια χρηματοδοτική δομή, είναι κάτι που είναι πολύ απαραίτητο. Κάτι σημαντικό για την αξιολόγηση συστημικών κινδύνων είναι να προσμετρήσουμε το βαθμό να δούμε τι ποιοτικό, ποιο είναι ο ποιοτικό χαρακτήρα του συστήματο. Δηλαδή το σύστημα πώ μπορεί να αυξήσει τι διακυμάνσει και πώ μετά από χρονική περίοδο το σύστημα μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικέ ανόδου αυξήσει και καθόδου, ξεκινώντα από ένα μέτριο επίπεδο. Ένα γκλονισμό μέτριο να τον αυξάνει σαν ισχυτή δηλαδή. Αυτό η συστημική αστάθεια του συστήματο είναι κάτι πάρα πολύ περίπλοκο σαν έννοια, ζητά ανάλυση της διασύνδεσης μεταξύ των διαφόρων φαινομένων που υπάρχουν. Κακή συμπεριφορά. Και πώς γίνεται, πώς υπάρχει επίδεση μεταξύ των εκθέσεων. Και τι γίνεται με τη συνετή διαχείριση, τι γίνεται με τους κανόνες σχετικούς, λογιστικούς κανόνες και τι γίνεται με τους ε, φορείς εξονόμησης κλπ. Ένα σημαντικό τομέα λοιπόν είναι η αξιολόγηση του συστημικού κινδύνου στα πλαίσια των διασυνδέσεων μεταξύ των πιστοτικών ιδρυμάτων σαν σύνολο και από τη μια μεριά και της πραγματικής οικονομίας. Διότι μπορεί εδώ να αντανακλώνται οι πραγματικές ελλείψεις ισορροπίας στην πραγματική οικονομία. Επομένως, μπορεί να προκύψουν ολέθρια αποτελέσματα όπως φάνηκε και από την πρόσφατη εμπειρία της κρίσης. Επομένως, είναι απαραίτητο να υπάρξει και μία υγιής μακροοικονομική πολιτική ώστε να εξαλειφθούν οι ανισότητες, οι ελλείψεις ε, ισορροπίας, οι οποίες από μόνες τους μπορούν να οδηγήσουν σε μια ακαμψία και σε μια αστάθεια στην πραγματική οικονομία. Είναι δύσκολο ιδίως να αξιολογήσουμε τις πηγές συστημικού κινδύνου γιατί βασίζονται στην αλληλεπίδραση διαφορών στοιχείων στο σύστημα και επομένως είναι από την φύση τους, από τα γενοφάσκια τους, είναι πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να τις αντιληφθεί κανείς και να τις καταμετρήσει. Πολλές φορές ο κίνδυνος αυτός αναδύεται με έναν τρόπο ο οποίος είναι απότομος και μη γραμμικός και Μόνο με μη στάνταρ αναλύσεις μπορεί κανείς να κατανοήσει την πηγή αυτών των κίνδυνων. Ο τρόπος με τον οποίο διαδίδεται ο κίνδυνος πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να το μοντελοποιήσει κανείς και να το αντιμετωπίσει. Υπάρχουν συσχετισμοί και μεταξύ τμήματων της οικονομίας που δεν είναι προφανείς και επομένως είναι απαραίτητο να ξέρουμε όχι μόνο τους διάβλους διαβίβασης αυτών των κινδύνων αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε και ότι είναι εύρωστο και ανθεκτικό το ίδιο το σύστημα. Συνήθως οι αναλυτές μπορούν να βασίζονται σε έγκαιρες και πρώιμες μορφές προειδοποίησης για δείκτες συστημικής σημασίας, όταν αυτοί οι δείκτες προσεγγίζουν ένα επίπεδο κινδύνου, αλλά για την ε, αξιολόγηση της ανθεκτικότητας του συστήματος μακροοικονομικά, μακροοικονομικές δοκιμασίες είναι απαραίτητες, μπορούν να εξασφαλίσουν εξάλλου και την ιεράρχηση των κινδύνων και να μπορούν να, θα μπορούσαν να οδηγήσουν και στην ανάπτυξη συστάσεων σε επίπεδο πολιτικής. Οι κεντρικές τράπεζες και οι ρυθμιστικοί φορείς σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να αναπτύξουν περαιτέρω αυτά τα εργαλεία και κατά την άποψή μου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, το ESRB, μπορεί να κάνει μια σημαντική συμβολή για να προωθήσει την ανάλυση του συστημικού κινδύνου, να συντονίσει τι αναλυτικές έρευνες και προσπάθειες και να συντονίσει τις ε, προσπάθειες που γινόνται από τι κεντρικέ τράπεζες και του ρυθμιστέ από όλα τα κράτη-μέλη. Εγώ πιστεύω επίση ότι ο λόγος αυτού του Συμβουλίου για την ανάλυση κινδύνου όσον αφορά την μετατροπή της ανάλυσης κινδύνου σε πρώιμες προειδοποιήσει και συγκεκριμένε συστάσεις για την πολιτική, καθώς και η ιεράρχηση του κινδύνου, θα μπορέσει να συμβάλλει ιδιαίτερα στο να είναι πιο ανθεκτικό το χρηματοοικονομικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι στο οποίο προσβλέπουμε όλοι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τρισέ. Προχωρούμε τώρα στις ερωτήσεις που θέτουν οι βουλευτές. Έχω εδώ ένα κατάλογο του ποιος θα θέσει ερώτημα από ποια πολιτική ομάδα. Θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι έχουμε το εξή σχήμα 1,5 λεπτό για κάθε ερωτώντα και στη συνέχεια λαμβάνει το λόγο ο κύριος Τρίσε ο οποίος απαντά σε ένα χρονικό διάστημα μέχρι τρία λεπτά. Ο κύριος Μπάλτς από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα εισαγωγική σας ομιλία. Έχω τρεις σύντομες ερωτήσεις λόγω πίεσης και χρόνου. Καταρχήν η στρατηγική εξόδου, την οποία αναφερθήκατε, και τα έκτακτα μέτρα, είπατε ότι θεωρείτε ότι πρέπει να αφαιρεθεί σε κάποιο σημείο η υπερβολική ρευστότητα στην αγορά. Θα ήθελα να ξέρω αν αυτό θα γίνει σε συμφωνία με τους εθνικούς υπουργούς, τα Εθνικά Υπουργεία Οικονομίας, που φυσικά έχουν τους εθνικά προγράμματα και κάνουν κινήσεις οι οποίες βασίζονται στα εθνικά τους προγράμματα. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πώς θα συνδυαστεί η δράση σας με αυτή των εθνικών υπουργείων. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα μη στάνταρ μέτρα, αναφερθήκατε σε ορισμένους κινδύνους που βλέπετε εσείς ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε ποιο βαθμό έχετε εσείς αξιολογήσει αυτούς τους κινδύνους, πόσο τακτικά τους αξιολογείτε και κατά πόσο υπάρχει μια συνεχής παρακολούθηση αυτών των κινδύνων. Και το δεύτερο κομμάτι της ίδιας σας ερώτησης είναι το εξής. Αν και όταν οι τράπεζες αφαιρέσουν αυτά τα τοξικά στοιχεία του ενεργητικού από τους ε, ισολογισμούς τους, εσείς θα ζητήσετε αυτό να γίνει τώρα ή να γίνει σε ένα μεταγενέστερο σημείο στον χρόνο. Τρίτον, μη είπατε ότι σε ορισμένου τομεί υπάρχει το λεγόμενο credit crunch, υπάρχει δηλαδή μια έλλειψη ρευστότητα και πιστώσεων. Όταν επανέλθει τώρα η εμπιστοσύνη στην αγορά και ξεκινήσει και η οικονομική ανάκαμψη, εξακολουθούν κατά την άποψή σας να υπάρχουν στενοποί σε ό,τι αφορά την παροχή πιστώσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην, κρίση και θα εμποδίσει κάποιες τράπεζες να δίνουν τις απαραίτητες πιστώσεις. Και εδώ πόσο συμφωνείτε με την τρίτη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ε, τράπεζα η οποία ζήτησε να υπάρξουν και νέε βραχυπρόθεσμες δράσεις για την εξασφάλιση της ρευστότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχει ένα ρολόι το οποίο όμως δεν λειτουργεί για τον χρόνο, θα το διορθώσουμε. Δεν θα εκμεταλλευτώ το γεγονός ότι δεν λειτουργεί το ρολόι, λέει ο κύριο Τρίσε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το ερώτημά σας. Θέλω να πω ότι σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη σταδιακή και έγκαιρη κατάργηση των ε, εκτάκτων μέτρων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυτά τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί για να είναι αυτοανερούμενα εν καιρό. Και φυσικά παρακολουθούμε από κοντά το τι συμβαίνει στην ίδια την αγορά και είναι σαφές ότι η κατάσταση της αγοράς όταν εισαγάγουμε για πρώτη φορά αυτά τα, τα μέτρα μετά από την κατάρρευση της Lehman Brothers η κατάσταση σήμερα είναι πολύ διαφορετική από την κατάσταση που επικρατούσε πριν από ένα χρόνο με την κατάρρευση των Lehman Brothers. Γι' αυτό έχουμε λάβει μια σειρά αποφάσεων για την ε, νέα στρατηγική που θα ακολουθήσουμε. Πάντα λέμε ότι θέλουμε να υπάρχει μια έγκαιρη αλλά σταδιακή αντιμετώπιση για να εξαλειφθούν εν καιρό τα μη στάνταρ αυτά μέτρα ώστε να λειτουργεί η αγορά ορθώς και φυσικά τώρα η αγορά ήδη λειτουργεί πολύ καλύτερα και οι φορείς σε εθνικό επίπεδο οι εθνικές αρχές έχουν πολύ καλή κατανόηση του τι πράττουμε. Έχουν και οι ίδιες αυτές οι εθνικές οικονομικές αρχές αντίστοιχα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντήσουν με ένα διαφορετικό τρόπο γιατί φυσικά αυτό εξαρτάται από την ε, χώρα στην οποία βρίσκονται. Σε ορισμένε χώρε η κατάσταση του χρηματοοικονομικού τομέα ήταν ιδιαίτερα οξία και δύσκολη. Σε άλλε χώρε δεν υπήρξε τόσο μεγάλη επιρροή τη κρίση. Υπήρξαν από όλους κινήσεις προσαρμογών. Εγώ προς το παρόν όμως δεν διαβλέπω κανένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά το συντονισμό με τις εθνικές αρχές, το οποίο ήταν το πρώτο σας ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημά σας τώρα. Θα σας έλεγα ότι προφανώς εξετάζουμε πολύ προσεκτικά την κατάσταση συνολικά και όπως ανέφερα στην εισαγωγική μου παρατήρηση, στην εισαγωγική μου ομιλία, Εμείς δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα παροχής πιστώσεων, κάποιο σημαντικό ε, πρόβλημα. Ξέρουμε ότι υπάρχει κάποια συρρήκνωση των πιστώσεων, ιδίως για, τα, για τις πιστώσεις οι οποίες είναι πιο βραχυπρόθεσμες, με ε, χρονικό διάστημα αποπληρωμής κάτω από πέντε χρόνια για τις πιστώσεις που είναι πιο μακροχρόνιες δεν υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα. Βλέπουμε γενικά συνολικά να υπάρχει μείωση των πιστώσεων οι οποίες έχουν δοθεί στον ε, τομέα των επιχειρήσεων αλλά εξακολουθούμε να παρακολουθούμε από πολύ κοντά αυτή τη διαδικασία για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει και βλέπουμε ότι προφανώς και η ζήτηση πιστώσεων έχει μειωθεί όπως συμβαίνει πάντα μετά από την εκκίνηση μιας οικονομικής ύφεσης εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στην ε, ύφεση. Δεν ήταν μια τεράστια, τεράστια έκταση ύφεση, αλλά έχει μειωθεί παρόλα αυτά σημαντικά η ζήτηση για πιστώσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο πάντα παρουσιάζεται σε τέτοιες χαμηλές φάσεις του οικονομικού κύκλου. Από τη δική μας λοιπόν πλευρά και μετά από την προσεκτική ανάλυση στην οποία έχουμε προβεί για την κατάσταση, βλέπουμε ότι ο κύριος καθοριστικός παράγων είναι η ζήτηση για επενδύσεις και όχι η προσφορά για τις επενδύσεις. Το τελευταίο σας ερώτημα τώρα, το κατά πόσο θα μπορούσαν να υπάρξουν και περαιτέρω κλειδονισμοί και μείζονες δυσκολίες, πρέπει να σας πω ναι, μπορούμε να περιμένουμε κάτι τέτοιο, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε επάγρυπνοι. Εξακολουθούμε να είμαστε σε μια κατάσταση η οποία απαιτεί επαγρύπνηση μια κατάσταση όπου εξακολουθούν να υπάρχουν αστάθμητα στοιχεία και αβεβαιότητες ακόμα στον οικονομικό χώρο. Υπάρχει ένα συστηματικό στοιχείο αβεβαιότητας, το οποίο λοιπόν πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καράς. Πάλι δεν δουλεύει αυτό το μαραθέτη το ρολόι. Θα χρησιμοποιήσουμε το σύστημα των κυτρίνων και των κοκκίνων καρτών. Ο κύριος Καράς, μία πάρα πολύ σύντομη ερώτηση. Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε της Τρισέ, την προηγούμενη εβδομάδα το Συμβούλιο πήρε μια απόφαση σε σχέση με την ε, ε, εποπτεία της Ευρωπαϊκής Χρηματαγοράς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανεξάρτητα από παράταξη αντέδρασε και είπε ότι δεν το ικανοποιεί αυτή η πρόταση, αυτή η απόφαση του Συμβουλίου. Ποια είναι τώρα η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Δεύτερον, ε, και θεωρούμε ότι η απόφαση του Συμβουλίου δεν καλύπτει την απαραίτητη εποπτεία των χρηματοοικονομικών αγορών. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Πρόκειται για το θέμα του λόγου μόχλευσης οι Αμερικανοί έχουν εισαγάγει ένα νέο, ένα νέο ορισμό για τη μόχλευση. Εσείς τι ακριβώς, ποια στοιχεία θα λάβετε για να υπολογίζετε το, τον λόγο μόχλευσης. Και το τρίτο ερώτημα, υπάρχουν χώρες όπως η Ελλάδα που έχει φτάσει ένα έλλειμμα της τάξης του 12%. Πώς εσείς μπορείτε να αντιμετωπίσετε ελλείμματα αυτού του ύψους στην περίπτωση, στην περίπτωση χωρών που ανήκουν στο ευρώ, στη ζώνη του ευρώ. Για το πρώτο σας ερώτημα. Είναι ένα πολύ ευρύ ερώτημα βεβαίως, γιατί ζητάτε την άποψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, όσον αφορά το πακέτο εποπτείας το οποίο έχει προβλέψει το Συμβούλιο. Θα έλεγα ότι σε αυτή τη φάση βεβαίως καταλαβαίνω ότι είναι ένα θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να πω το εξή. Όπως γνωρίζετε, δεν είναι ό,τι καλύτερο, δεν είναι η πρώτη μας επιλογή. Αλλά δεδομένου του περίπλοκου της κατάστασης και της ευαισθησίας ε, των διαφόρων κυβερνήσεων ε, των 27 κρατών μελών, θα έλεγα ότι η Σουηδική Προεδρία έκανε καλή δουλειά. Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη μας επιλογή, αλλά από την άλλη το αποτέλεσμα είναι αρκετά αξιόλογο, λαμβανομένης υπόψη βέβαια της ε, δυσκολίας ε, και των διαφορετικών ευαισθησιών που υπάρχουν στο πλαίσιο των ε, εκτελεστικών ε, φορέων. Όσον αφορά τώρα το λόγο μόχλευσης, γνωρίζετε ότι Υπάρχει έντονη συζήτηση στο πλαίσιο της ομάδας της Βασιλείας και γνωρίζετε τι διδάγματα πρέπει να πάρουμε βέβαια από την ε, τρέχουσα κρίση. Η ιδέα ότι πρέπει να αποφύγουμε την προκυκλικότητα και ότι πρέπει να δουλέψουμε για να το πετύχουμε αυτό είναι μια πολύ καλή οδός για να πετύχουμε την αύξηση του δυναμικού ε, του τραπεζικού τομέα. Έχουμε βέβαια και τις ε, διάφορες ε, απαιτήσεις για τη ροή των κεφαλαίων ε, που πρέπει να τις συσχετίσουμε με, το, με τους κινδύνους που δεν ήταν βέβαια η περίπτωση με τη Βασιλεία 1, αν ξεχάσουμε για παράδειγμα τους κινδύνους που ήταν ενσωματωμένοι στο θέμα, στην όλη διαδικασία των χρεογράφων, αλλά η ιδέα του να έχουμε ένα λόγο μόχλευσης έχει συζητηθεί και η Επιτροπή της Βασιλείας εξακολουθεί να ε, το να επεξεργάζεται, να επεξεργάζεται αυτή τη δυνατότητα. Δεν θα πρέπει να είναι βέβαια ένας λόγος ο οποίος πιστεύω ότι πρέπει πρώτα να βλέπουμε το βασικό κίνδυνο που υπάρχει, αλλά ως ε, δεύτερη επιλογή να μην ε, υπάρχει, για να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τα πράγματα, θα μπορούσε να υπάρχει ένας λόγος μόχλευσης και αυτό έχει συζητηθεί ε, στην Επιτροπή Βασιλείας Το τρίτο θέμα που θέσατε Το ένα αφορά ε, το, τη, τη, το εκτός της Ευρωζώνης ε, και εντός ε, της Ευρωζώνης. Η κατάσταση βέβαια στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πράγματι γνωρίζουμε όλοι τα αριθμητικά στοιχεία και γνωρίζουμε τις πολύ γενναίες αποφάσεις που θα πρέπει να λάβουμε για να μπορέσει να βελτιωθεί η κατάσταση της ε, φορολογικής πολιτικής, για παράδειγμα, ολόκληρη τη στρατηγική επίσης της χώρας. Επομένως, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, χρειάζονται πολύ γενναίες αποφάσεις, αλλά και είναι πολύ απαραίτητα αυτά τα μέτρα και είμαι πεπισμένο ότι η κυβέρνηση της ε, κυβέρνησης ε, θα έχει τη διορατικότητα να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Είναι λίγο άδικο να δίνετε απάντηση σε τρία λεπτά όταν τρει ερωτήσει σα υποβάλλονται και στο τέλο δεν θα μπορέσουν όλοι να πάρουν το λόγο. Κύριο Φέρμπερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τρισέ, υπάρχουν κάποια σημάδια ότι οι τράπεζες έχουν δείξει την, τάξη, την τάση να χρησιμοποιούν πιστώσεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για κερδοσκοπικούς λόγους και έτσι μπορεί να δημιουργηθεί μια νέα φυσαλίδα. Έχουμε ήδη αντιμετωπίσει το θέμα της ε, έλλειψης, πιστο... έλλειψης ρευστότητος. Δεν ξέρω λοιπόν αν θα τροφοδοτήσει μια νέα κερδοσκοπική φυσαλίδα η φτηνή ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θέλετε λοιπόν να την περιορίσετε, θα κάνετε τα απαραίτητα για, για κάτι τέτοιο. Πώς γίνεται λοιπόν όλα αυτά τα, όλη αυτή η φτηνή ρευστότητα την οποία εσείς θέτετε στην ε, διάθεση των τραπεζών να μην καταλήγει στις επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να χρηματοδοτούν. Είναι απλό το ερώτημα και μπορείτε να απαντήσετε εν συντομία. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό είναι σημαντικότατο ζήτημα. Πρέπει συνεχώς να σταθμίζουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα έλεγα και όλες οι αδελφές κεντρικές τράπεζες να σταθμίζουμε τους κινδύνους, τους σχετικούς που σχετίζονται με τα μέτρα που πήραμε, τα έκτακτα μέτρα, διότι ήμασταν εν μέσω της κρίσεως και το κίνδυνο που αναλαμβάναμε. Κατά πόσο θα εκπνεύσουν, θα λήξουν αυτά τα μέτρα πολύ νωρίς ή πολύ αργά. Και γι' αυτό είπα πολύ ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει αποδεκτή εκ των προτέρων τάσης πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν περισσότεροι κίνδυνοι που συνδέονται με πρώιμη έξοδο από ότι με καθυστερημένη έξοδο. Εκ των προτέρων λύση δεν μπορούμε να την προβλέψουμε να την εφαρμόσουμε. Η κατάσταση είναι τέτοια που πρέπει να βρούμε ακριβώς τη σωστή εξισορρόπηση των κινδύνων. Και είναι πολύ σχετικό το ερώτημά σας. Καταρχάς, γι' αυτό την περασμένη Πέμπτη πήραμε την απόφαση που πήραμε. Θεωρήσαμε ότι ήρθε η ώρα σταδιακά, προοδευτικά, έγκαιρα να ξεκινήσουμε την λήξη της σταδιακή αυτών των εκτάκτων μέτρων. Τούτων λεχθέντων ε, για τις τράπεζες έχουμε σαφέστατο μήνυμα. Λέμε στις τράπεζες. Ό,τι κάναμε, ό,τι κάνουμε δεν έγινε για τα όμορφα σας μάτια. Έγιναν διότι έχετε ρόλο βασικό να διαδραματίσετε στις οικονομίες της αγοράς. Πρέπει να αξιολογήσετε τους κινδύνους και να δανείσετε. Αυτή είναι η λειτουργία σας. Και ό,τι κάναμε, και τολμώ να πω ότι ό,τι έγινε από τις κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια, από τους φορολογουμένους, οι κίνδυνοι που ανελήφθησαν, όλα αυτά έγιναν με ακριβώς αυτό το σκοπό. Και για κανέναν άλλο λόγο, αυτό είναι σίγουρο. Είναι ισχυρότατο το μήνυμα του λεχθέντος να πω ότι η ανάλυση μας αυτή τη στιγμή δείχνει ότι βασικός λόγος για τα παρατηρούμενα όσον αφορά τις πιστώσεις ε, οφείλονται στη ζήτηση και όχι σε μη έλλειψη πιστώσεων, έλλειψη παροχής προμήθειας. Αλλά το μήνυμά μας είναι αυτό προς τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εκείνοι που θεωρούν ότι τίποτα δεν έγινε και τώρα όλα είναι κανονικά διότι ξαναλειτουργεί η αγορά πλανώνται πλάνη νικτράν αποφύγαμε την ύφεση διότι ήμασταν αρκετά τολμηροί και έγκαιρα πήραμε αυτά τα μέτρα που ανέφερα. Και όταν λέω πήραμε, εμεί, οι κεντρικέ τράπεζε εννοώ, και οι ίδιε ε, οι κυβερνήσεις. Και το να μην το καταλάβει κανεί αυτό είναι εσφαλμένο. Διότι τολμώ να πω ότι δεν εμπιστεύομαι το ότι ο φορολογούμενος δύο φορές θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που αντιμετωπίσαμε για να αντιμετωπίσουμε την ύφεση. Την ύφεση συγγνώμη. Άρα θέλουμε να λειτουργεί πολύ, με πολύ πιο ανθεκτικό τρόπο το σύστημα. Αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ερώτηση από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τρισέ, από τις προηγούμενες σας απαντήσεις, ε, αν κατάλαβα καλά, όσον αφορά την ε, αναστρεψιμότητα αυτών των πέντε εκτάκτων μέτρων. είπατε ότι είναι όλα αναστρέψιμα, αλλά ότι εξαρτάται από τη χρονική στιγμή. Δηλαδή ότι αν ε, τα διατηρήσουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με την κατάργησή τους. Το δεύτερο, η δεύτερη όμως έννοια της αναστεψιμότητας είναι η, τα ίδια τα μέτρα διεξόδου από την κρίση. Στη χειρότερη περίπτωση, για παράδειγμα, αν έχουμε αυτή τη στρατηγική εξόδου Μπορούμε να τη σταματήσουμε κάποια στιγμή. Υπάρχει κάποιο είδου ε, κεκτημένη ταχύτητα τέλο πάντων για... λόγω τη οποία δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε. Επίση, ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προφανώ δεν θα περιμένει τι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει ε, να καταρτήσουν τη δική του στρατηγική. Καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα σε σχέση με έναν ανεξάρτητο φορέα όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ε, υπάρχει μια δυσκολία, το καταλαβαίνω, αλλά βρίσκεται ε, ότι τα προβλήματα είναι σημαντικά. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, αυτή η ερώτηση είναι πολύ σημαντική. Όπως είπα, προσπαθούμε να αξιολογήσουμε την κατάλληλη στιγμή για να συνοδεύσουμε τη βελτίωση που παρατηρούμε στις ε, ε, χρηματοπιστωτικές αγορές, στις χρηματαγορές κυρίως, ε, για να λάβουμε την απαραίτητη απόφαση. Πρέπει όμως να υπάρξει μια εξισορρόμηση μεταξύ του κινδύνου να καθυστερήσουμε πάρα πολύ σε αυτή την σταδιακή κατάργηση των εκτάκτων μετρών. Είπα ότι δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη λύση που θα προτιμήσουμε, αλλά η άλλη παρατήρηση που κάνατε που πολύ σωστή ήταν, δηλαδή οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη μη κατάργηση που μπορεί ή μια κατάργηση που μπορεί να καθυστερήσει. Καταλαβαίνω, όντω υπάρχει κίνδυνο, υπάρχουν αγορέ που ενδεχομένω να εφιστούν σε αυτή τη διαδικασία και υπάρχει και το θέμα του αντιπαραγωγικού αντικτύπου που μπορεί να υπάρξει συνεπώ στην κερδοσκοπία ε, σε συγκεκριμένε αγορές με διάφορα ε, μέσα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έγκαιροι. Τώρα, σε ποιο επίπεδο θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να σας ε, αφήσουμε απ' έξω ή να ε, σταματήσουμε κάποια μέτρα. Εμείς έχουμε προβλέψει κατάργηση. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο αμφισβητείται αυτή τη στιγμή από τους παρατηρητές των αγορών, από την παρατήρηση των αγορών. Ελπίζω να μην βρεθούμε παγιδευμένοι σε μια κατάσταση τέτοια. Βέβαια είναι απρόβλεπτα τα πράγματα ε, για το μέλλον και υπάρχει κάποιο είδους αβεβαιότητα ακόμη, αλλά προσπαθούσαμε να έχουμε μια κάπως αντικειμενική παρατήρηση των ε, χρηματοπιστωτικών αγορών, αλλά η άποψή μου είναι ότι δεν θα σταματήσετε να συμμετέχετε και το λέω αυτό λόγω της ε, φύσεως των μη συμβατικών μέτρων που έχουμε λάβει όσον αφορά τις κυβερνήσεις. Ας το δούμε πρακτικά. Τι γίνεται. Σε ορισμένες περιπτώσεις ε, ήδη έχουν καταργηθεί κάποια μέτρα σε πολλές χώρες. Ε, οι εμπορικές τράπεζες ε, ήδη ξεπληρώνουν το κυβερνητικό χρέος τους ή οποιαδήποτε βοήθεια τους δόθηκε σε μετοχές. Ε, οπότε βλέπετε σιγά σιγά ότι το γεγονός ότι συμπεριφέρεται πολύ καλύτερα η αγορά κατά κάποιο τρόπο από μόνο του σταματά τα μέτρα τα οποία έχουν ε, ληφθεί σε πολλές περιπτώσεις. Ε, οι εγγυήσει ε, για μεσοπρόθεσμη αναχρηματοδότηση που είχαν προβλεφθεί για πολλές τράπεζες έχει, δεν, δεν χρησιμοποιείται πλέον γιατί οι αγορές συμπεριφέρονται καλύτερα. Ενδεχομένως λοιπόν ορισμένα μέτρα να πάβουν να υφίστανται για πολύ για λόγους ε, φυσιολογικής εξέλιξης. Ε, υπήρξε κάποια υποστήριξη, αλλά δεν χρειάζεται πλέον. Και αυτό είναι κάτι καλό βεβαίως. Θα είναι πολύ κακό να συνεχίσουμε να παρέχουμε ε, στήριξη η οποία πλέον δεν χρειάζεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η άλλη Μακάρθη. Πατρίτσια, να επιστρέψω σε αυτό το θέμα. για το, Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Πώς θα υπάρξει στενή συνεργασία με αυτό όσον αφορά την αρνητική δουλειά και την έρευνα που γίνεται και πώς θα αναλύονται οι πληροφορίες που θα συλλέγονται. Θα ήθελα να ξέρω πώς θα λειτουργήσει η συστημική ανάλυση. Ξεκίνησε ένα πρόγραμμα συλλογής στοιχείων, συλλογής γνώσεων για το συστημικό κίνδυνο. Για την προετοιμασία της κεντρικής προσπάθειας. Τι συνεπάγεται αυτό, πώς έχετε προχωρήσει, ποιος κάνει τη δουλειά, ε, γίνεται εντό τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή όχι. Έχετε κάποια πρώτα μαθήματα που μπορείτε να αντλήσετε από τη δουλειά που κάνατε μέχρι τώρα. Ξεκίνησε η διαδικασία προσλήψεων ήδη για εκείνου που θα εργαστούν στον τομέα αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα αρκετά θέματα για να απαντήσετε εντό τριλέπτου. Ευχαριστώ, λέει ο κύριο Τρισέ. Πρώτα απ' όλα, η όδια έννοια για το Συμβούλιο αυτός Αναλύσεως Συστημικού Κινδυνού ήταν για να υπάρχει στενή ε, συνεργασία, μάλλον και τα ΚΕΤΑΠΕΣ να συνεργάζεται με, αυτή την, με το Φορέα Αναλύσεως Συστημικού Κινδύνου. Και τα μέλη έχουν ε, δικαίωμα ψήφου και αυτό το Συμβούλιο συνεργάζεται στενά με τον υπεύθυνο για τον μακροοικονομικό έλεγχο. Πρέπει λοιπόν όλες οι πληροφορίες που είναι στα χέρια όλων των συμμετεχόντων στο εγχείρημα, κεντρική τράπεζα δηλαδή, και ελεγκτικές αρχές και ελεγκτικές αρχές, υποπτικές αρχές σε εθνικό επίπεδο να λειτουργούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι ίδιες οι κεντρικές τράπεζες θέλουν να συμμετάσχουν με το πιο επαγγελματικό τρόπο στην προσπάθεια. Ούτως ώστε όχι να μην συγκεντρωθούμε επί των μικροελέγχων σε μικροοικονομικό επίπεδο και να υπάρχει σαφής κατανομή των ευθυνών και να μπορέσουμε να επικεντρωθούμε επί του συστημικού ελέγχου όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών και ανταλλαγή γνώσεων, ναι. Επεξεργαζόμαστε τη χρηματοδοτική σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στις, ευρωπαϊκές, και στις κεντρικές τράπεζες των χωρών. Είναι σημαντική ευθύνη που υπέχουμε επειδή οι κεντρικές τράπεζες ενδιαφέρονται μέσω μακροπρόθεσμα για διάφορα θέματα, επιθυμούν σταθερότητα, τιμών και χρηματοπιστατική σταθερότητα και επειδή είναι ανεξάρτητες οι κεντρικές τράπεζες, θεωρήθηκε ως ενδεδειγμένο να τους δώσουμε αυτή την ευθύνη αξιολογήσεως του συστημικού κινδύνου, συνεχούς αξιολογήσεως, χωρίς όμως αυτές οι τράπεζες να αντικαθιστούν ιονδήποτε θεσμό και χωρίς να υπάρχει σύγχυση καθηκόντων. Ερευνούμε όλες τις πτυχές, θεωρητικές και πρακτικές. Χρειάζεται πολλή δουλειά. Και σε όλο τον κόσμο ιδιαίτερα στην Ευρώπη βέβαια, διότι έχουμε και φιλοδοξίες. Θέλουμε να έχουμε ενιαία αγορά που λειτουργεί όσο καλύτερα γίνεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σε επίπεδο 27 κρατών μελών κινούμεθα όσον αφορά το Συμβούλιο αυτό για την ανάλυση του κινδύνου και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξεκίνησε η διαδικασία χρήσεως της υφιστάμενης γνώσεως να χρησιμοποιήσουμε το ειδικευμένο προσωπικό που υπάρχει στις διάφορες κεντρικές τράπεζες, στις 27 κεντρικές τράπεζες, ούτω ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν χρησιμοποιούμε μόνο τους δικούς μας πόρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τις δικές μας γνώσεις και την χρήση του ανθρωπίνου κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά κινηθούμε ευρύτερα. Πιο σφαιρικά. Και το Κοινοβούλιο από την αρχή επιθυμούσε κάτι τέτοιο, το γνωρίζω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Σίλβη, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε στη συνεδρία της Επιτροπής μας. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της εποπτείας. Απαντήσατε στον κύριο Καράς, ο οποίος εξέφρασε μια απόψη που νομίζω ότι την συμμεριζόμαστε οι περισσότεροι από εμά και είναι φιλόδοξη από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προς ποια κατεύθυνση θα πήγαινε η πρώτη σας επιλογή για τα θέματα αυτά και στις ε, εργασίες που θα κάνει τώρα το Κοινοβούλιο εφόσον το, κοινοβούλιο, το Συμβούλιο έχει δώσει τη δική του άποψη για τα θέματα αυτά, για σας ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να τύχουν προτεραιότητας για να ενισχυθούν οι εποπτικοί φορείς, <clears throat> δεδομένου ότι όπως είπατε και όπως είπαμε και εμείς, είναι απαραίτητο να δοθεί το μήνυμα στον πληθυσμό της Ευρώπης ότι δεν βρισκόμαστε σε σενάριο business as usual, ότι θέλουμε πραγματικά ένα σύστημα το οποίο θα ελέγχει και θα αποτρέπει τους κινδύνους. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνοψίσω το τι, σε τι συνίσταται η πρώτη μου επιλογή με τον πιο απλό δυνατό τρόπο σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πάντα η θέση μας ήταν ότι μια κεντρική τράπεζα πρέπει να είναι πολύ κοντά στην μικροεποπτεία και αυτό είναι μια καλύτερη αντίληψη από μια κεντρική τράπεζα η οποία δεν επεμβαίνει καθόλου σε επίπεδο εποπτείας σε μικροοικονομικό επίπεδο. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουν επιζητήσει οι διευθυντές της Κεντρικής Τράπεζας πολύ πριν από την κρίση και το έχουμε διαδηλώσει δημόσια ότι αυτή ήταν η θέση μας. Να υποστήριξουμε τη μικροοικονομική εποπτεία. Όταν μας έθεσε το ερώτημα αυτό η Επιτροπή Ντελαροζιέρ, εμείς είχαμε πει ότι είμαστε έτοιμοι ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εάν αυτό ήταν απαραίτητο, να παίξουμε ένα διαιτητικό ρόλο μεταξύ της μικροοικονομικής εποπτείας των τραπεζών, των φορέων των πιστοτικών που είχαν, επίσης διαμεθοριακό χαρακτήρα και επέκεινα τη ζώνη του ευρώ. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως κεντρική τράπεζα της ζώνης του ευρώ, όχι βέβαια ως φορέας που έχει ένα ρόλο σε επίπεδο 27 χωρών, θα μπορούσε να έχει αυτόν τον υποπτικό ρόλο. Αυτό δεν το δέχτηκε η Επιτροπή Ντέλα και προφανώς όπως γνωρίζετε καλύτερα για από μένα φυσικά δεν το απεδέχθη ούτε το Συμβούλιο ούτε η Κομισιόν. Το λέω αυτό παρενθετικά. Η δεύτερη καλύτερη επιλογή που θα είχαμε διατηρήσει αν ήταν δυνατόν ήταν το να μπορούμε σε επίπεδο εποπτικών φορέων, εάν αυτό είναι απαραίτητο, να έχουμε περισσότερες ευθύνες και αρμοδιότητες ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Τώρα, είναι σαφές ότι αυτό το οποίο αποφασίστηκε από το Συμβούλιο δεν ανταποκρίνεται στην πρώτη επιλογή που θα είχε διατυπώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά φυσικά εγώ ελπίζω ότι η Σουηδική Προεδρία δεν θα μπορούσε, ε, πιστεύω ότι η Σουηδική Προεδρία θα μπορούσε να κάνει κάτι πολύ καλύτερο τη στιγμή που ήταν σαφής η αντίθεση άλλων κρατών. Ο κ. Καράς χωρίς μικρόφωνο. Γνωρίζω ότι το Κοινοβούλιο έχει το κλειδί ίσω της λύσης. Γι' αυτό εγώ απαντώ στο ερώτημά σα για το ποια είναι η πρώτη προτεραιότητα που θα είχα εγώ και ποια θα ήταν η καλύτερη λύση για μένα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την εποπτεία σε μικροοικονομικό επίπεδο. Και το ερώτημά σας, ελπίζω ότι σας απήντησα κυρία Γκουλάρα. Ναι. Ευχαριστώ, λέει Ευχαριστώ. Αν μπορείτε κύριε Τρισέ, μπορείτε να σχολιάσετε τη δύναμη του ευρώ τη σημερινή έναντι των άλλων ε, νομισμάτων, κυρίω έναντι των άλλων σημαντικών χωρών προ τι οποίε εξάγει η Ευρωζώνη. Κάναμε κρόα την περασμένη εβδομάδα και εκεί τονίστηκε ότι το σουηδικό μοντέλο ήταν επιτυχέ στι αρχέ τη δεκαετία του 90 μόνο αφού υποτιμήθηκε η σουηδική κορώνα και μετά είχαμε μια δεκαετία πολύ ε, αναπτύξεω μεγάλη των εξαγωγών. Βλέποντα την ισχύ που έχει το ευρώ, τη δύναμη που έχει το ευρώ σήμερα, μειώνεται η δυνατότητα εξαγωγών. Μήπω αυτό δημιουργεί προβλήματα, έχετε κάποιο σχόλιο όσον αφορά την δύναμη που έχει το ευρώ, την, αξία που έχει το ευρώ. Συναρτήσει των άλλων νομισμάτων. Ευχαριστώ κυρία μου, λέει και ο Στρισέ. Υπάρχουν δύο ερωτήσεις που ετέθησαν. Σχόλιο και ερώτημα θέσατε. Το ευρώ καταρχάς έναντι των άλλων σημαντικών νομισμάτων ισοτιμίας και μετά η λειτουργία της ίδια ενιαία αγοράς των 27 χωρών δηλαδή με τα διάφορα νομίσματα. Όσον αφορά τη θέση του ευρώ, που είναι ένα από τα σημαντικά νομίσματα. Ξέρω ότι θεωρείται κάτι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το ότι οι αρχές των ΗΠΑ επιθυμούν να επαναλαμβάνουν ότι το ισχυρό δολάριο είναι προς όφελος των Ηνωμένων Πολιτειών και προς όφελος των εταίρων των Ηνωμένων Πολιτειών θα έλεγα. Εντές των διαφόρων διακειμενόμενων νομισμάτων και ισοτιμιών. Κάτι πολύ σημαντικό για την ευμάρεια της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθερότητά της. Τώρα η θέση του ευρώ που είναι ένα από τα σημαντικά νομίσματα. Θα έλεγα ότι αφορά τα μη διακειμενόμενα νομίσματα που δεν διακειμένονται σε παγκόσμιο επίπεδο κυρίως νομίσματα αναδειωμένων οικονομιών κυρίως της χωρών της Ασίας που βρίσκονται σε ένα επίπεδο που δεν αξιολογείται και επαρκώς και λόγω παρεμβάσεων θα έλεγα ότι σταδιακή και τακτική αξιολόγηση αυτών των των νομισμάτων έναντι ευρώ και έναντι δολαρίου, δηλαδή έναντι των βασικών νομισμάτων σε ελεύθερη διακύμανση, είναι κάτι προ όφελο τη παγκόσμια ευμάρεια και σταθερότητα. Τώρα εντό της ενιαίας αγοράς αναφέρει η συνθήκη όπως γνωρίζετε ότι ο συσχετισμός ισοτιμιών είναι κάτι προς κοινών όφελος και είναι σημαντικό καμία συγκεκριμένη χώρα να ισχυρίζεται ότι θέλει ένα νόμισμα να είναι όσο το δυνατόν πιο αδύναμο εντός της ενίας αγοράς των 27. Υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όμως καμιά χώρα, είμαι σίγουρος γι' αυτό, δεν προσπαθεί να βρεθεί σε πλεονεκτική θέση που εδράζεται επί μιας τέτοιας πολιτικής. Και τουλάχιστον δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια τέτοια περίσταση και πιο συγκεκριμένα δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο για την Σουηδία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε. Θα συνεχίσω στα αγγλικά και να απαντήσετε κι εσείς στα αγγλικά. Κάτι που μας απασχολεί πολύ και θα ήθελα και εγώ να ακούσω την ειλικρινή σας άποψη γι' αυτό, είναι κάτι το οποίο διαβάσαμε στον τύπο την ε, σχεδόν το σχεδόν φορολογικό ρόλο που έλαβε, που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το θέμα των collaterals, των εγγυήσεων, ειδικότερα για τίτλοι που βασίζονται για, τα, τίτλους που βασίζονται σε στοιχεία ενεργητικού. Ε, είπατε ότι δεν θέλετε να έχετε έκτακτα μέτρα πλέον και εμείς δεν θέλουμε να δούμε στρέβλωση των αγορών. Ενδεχομένως ε, δεν ξέρουμε αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να συνεχίσει να αναλαμβάνει αυτό το ε, ρόλο. Η δεύτερη μου ερώτηση είναι η εξής. Κατά την άποψή σας, κατά την εκτίμησή σας, πόσο μεγάλη είναι ακόμη η έκθεση των ε, χρηματοπιστωτικών ε, φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε κινδύνους το 2010 μισό τρισεκατομμύριο, ένα τρισεκατομμύριο, πόσο είναι κατά την άποψή σας. Thank you very much indeed. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την πρώτη σας ερώτηση, Πριν από την κρίση, όπως γνωρίζετε, πριν αρχίσει η κρίση, για μας δηλαδή στις 9 Αυγούστου 2007 όπου άρχισαν οι πρώτες, ε, άρχισε η πρώτη αναστάτωση, υπήρχε ένα πλαίσιο ενεχείρων που ήταν ε, ευρύτερο από ορισμένων εθνικών ε, τραπεζών δεχόμασταν ε, όχι μόνο τα κρατικά έγγραφα αλλά και τα ομόλογα αλλά και τα ιδιωτικά ομόλογα. Βέβαια από τότε έχουν υπάρξει πολύ μεγάλες αλλαγές. Αποφασίστηκε λόγω εν μέρη και της κρίσης να ε, δεχθούμε και τα ε, ιδιωτικά ομόλογα. Το γεγονός λοιπόν ότι δεχθήκαμε ε, το ABS αλλά και τα ε, ιδιωτικά δάνεια από την αρχή είναι κάτι το οποίο ε, ήταν σύμφωνο με αυτό που είχαμε φασίσει από την αρχή του ευρώ, όχι υποχρεωτικά στο πλαίσιο μιας κρίσης, απλώς στην κρίση ε, διευρύναμε ακόμη περισσότερο το πλαίσιο των ενεχείρων και επίσης είπαμε ότι παρακολουθούσαμε ε, πολύ στενά τους διάφορους κινδύνους και ενδεχομένως πρόσφατα να είδατε ότι λάβαμε αποφάσεις που δικαιολογούνται ακριβώς από το γεγονός ότι θέλαμε να ε, μειώσουμε τον κίνδυνο ε, στο πλαίσιο, στο πλαίσιο αυτό. Όσον αφορά τώρα την αξιολόγηση των ABS, ε, προσπαθούμε στο ίδιο το σύστημα να μειώσουμε τους κινδύνους. Νομίζουμε ότι είναι αρκετά, κατα... είναι αρκετά καλά τα πράγματα, αλλά μπορούμε ανα πάσα στιγμή βέβαια να προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο. Η τελευταία μας βελτίωση έχει, ε, ε έγινε πριν από μερικές ημέρες. Τώρα, ο, ο, όσον αφορά τις τράπεζες ε, ε, της Ευρωζώνης, τα νέα τα νέα μας μέτρα. Έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε ότι θα έπρεπε να είμαστε κάπως προσεκτικοί γιατί όντως ε, παρουσιάστηκαν κάποια ε, στοιχεία ε, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έκανε το ίδιο. Εμείς είμαστε πολύ προσεκτικοί. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει μειώσει το δικό του επίπεδο αξιολόγησης, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί οι τράπεζες δεν είναι στην ίδια κατάσταση όλες. Υπάρχουν τράπεζες που είναι σε πολύ καλή κατάσταση, που είναι πολύ προσεκτικές και άλλες που δεν είναι. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα προηγούμενα ε, ε, οι προηγούμενες αξίες ενεργητικού δεν είναι πλέον πρόβλημα ε, αν σκεφτούμε δηλαδή τι συνέβαινε στο παρελθόν, το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι υπήρξε μια πολύ έντονη ύφεση, έχουν βελτιωθεί τα πράγματα αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια προβλήματα και υπάρχουν ε, πιστώσεις που θα χρειαστούν θα χρειαστούν ε, ε, την αποδοχή ζημιών, η διαγραφή των ζημιών. Τώρα, το κέρδος ε, που αναμένουμε μέχρι για παράδειγμα το τέλος του επόμενου έτους θα είναι ανάλογα με ε, τα νέες, με τις διαγραφές απολειών ε, που, μπορούν, που μπορεί να συμβούν μετά το τέλος της ύφεσης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κουντής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Τρισέ, με τον τρόπο που έχει θεσπιστεί η ονέ και το ευρώ δεν προβλέπεται δανεισμός, μηχανισμός δανεισμού τελευταίας καταφυγής για μια χώρα που αντιμετωπίζει προβλήματα ή υφίσταται κερδοσκοπικά παιχνίδια. Όταν μια χώρα δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί σε μια τέτοια περίπτωση είτε να εκδώσει νέο χρήμα, είτε να καταφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όταν μια χώρα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι στη ζώνη του ευρώ, όπως άκουσα και είπατε σήμερα, αν καλά άκουσα, προβλέπεται μηχανισμός δανεισμού. Όμως, σε μια χώρα που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι στη ζώνη του ευρώ, όπως η Ελλάδα, δεν προβλέπεται τέτοιος μηχανισμός δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τι γίνεται λοιπόν, οι εμπορικές ελληνικές τράπεζες δανείζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με επιτόκιο 1%, στη συνέχεια δανείζουν το δημόσιο με επιτόκιο 4% και καταλαβαίνετε ότι είναι μια επένδυση χωρίς ρίσκο που φτάνει στα όρια της κερδοσκοπία. Η κατάσταση δημιουργεί αδιέξοδα με κερδισμένους τις εμπορικές τράπεζες και χαμένη την πραγματική οικονομία που δεν έχει εισπράξει ακόμα τη ρευστότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κατόπιν τούτου σας ερωτώ κύριε Τρισέ, πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και επειδή αναφερθήκατε στην περίπτωση της Ελλάδας, τι εννοείτε να ληφθούν γενναίες αποφάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έλεγα πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι χώρες της ζώνης του ευρώ ότι οι χώρες αυτές λοιπόν δεν είναι επιλέξιμες για ορισμένα έκτακτα μέτρα όπως αυτό που αναφέρατε, δηλαδή η προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η ενίσχυση στο ισοζύγιο πληρωμών που να προέρχεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση η παρουσία στη ζώνη του ευρώ, η συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ σημαίνει ότι το τρέχον ε, ισοζύγιο πληρωμών θα πρέπει να χρηματοδοτείται αυτόματα μέσα στην ε, ζώνη του ευρώ. Αυτό λοιπόν είναι ένα όφελος το οποίο αποκομίζει κανείς από την ίδια τη συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ. Αφ' αυτού αυτό είναι μια τεράστια βοήθεια λοιπόν είναι ένα είδος έμεσης αλλά πολύ σημαντικής αλληλεγγύης η οποία υφίσταται μεταξύ όλων των χωρών που ανήκουν στην ίδια περιοχή ενιαίου νομίσματος. Και αυτό το όφελος ήταν πολύ φανερό τους τελευταίους μήνες. Τώρα σε ό,τι αφορά τα απαραίτητα μέτρα, τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν, νομίζω ότι αυτά καθορίζονται από τις ίδιες τις συνθήκες τις οποίες διέρχεται η Ελλάδα. Και δεν αφορούν μια συγκεκριμένη χώρα και μόνο τα μέτρα αυτά. Εσείς αναφέραστε σε μια συγκεκριμένη χώρα. Εγώ θα έλεγα ότι όλες οι χώρες συλλήβδιν της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στα νοικοκυριά εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις, είτε είναι οι επιχειρήσει πιστοτικού χαρακτήρα ή όχι, ότι υπάρχει μια βιώσιμη στρατηγική σε ό,τι αφορά την εξυγίανση των ε, δημοσίων οικονομικών. Χωρίς όλα αυτά δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ούτε από τους καταναλωτές και τα νοικοκύρα, ούτε και από τους επιχειρηματίες. Πώς θα μπορέσετε να έχετε μια οικονομική ανάκαμψη, ελήψη εμπιστοσύνη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Προφανώς έχει και κάποιο ρόλο το τίμημα της αναχρηματοδότησης για το εθνικό θησαυροφυλάκιο. Όταν δεν υπάρχει μια αξιόπιστη στρατηγική μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στο δημοσιονομικό τομέα, πώς μπορείτε να μειώσετε το spread, διότι η αγορά δεν έχει κανένα λόγο να έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από ότι οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά σε μια χώρα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι προκύπτουν πολλές δυσκολίες, διότι είναι πολύ πιο επαχθές και πολυδάπανο το να αναχρηματοδοτεί κανείς τους κρατικούς πόρους. <clears throat> Πολύ σωστά λοιπόν λέτε ότι το καλύτερο σημάδι είναι ακριβώς το καλύτερο σημάδι της οικονομικής ανάκαμψης κατά κάποιο τρόπο, ακόμα και αν υπάρχουν προβλήματα. Όλοι βασίζονται στο επίπεδο στο επιτόκιο αναχρηματοδότησης των κρατικών πόρων, δηλαδή στο spread. Αυτό ακριβώ. Όλοι οι άλλοι φορεί αναχρηματοδοτούνται σε υψηλότερα επιτόκια. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί να υπάρξει δράση σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Ο Χάνς Πέτερ Μάρτιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία αναφέρατε και αναφερθήκατε σε όλες τις περιοχές του κόσμου σχεδόν. Για την Ελλάδα έχετε πει δύο φορές ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη. Τι σημαίνει αυτό όμως, μπορείτε να είστε λίγο πιο σαφείς. Θα φτάνατε στο σημείο να πείτε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρξει μια εξέλιξη στην Ελλάδα όπως αυτή στην Αργεντινή πριν από 10 χρόνια. Θα μπορούσατε να φανταστείτε η Ελλάδα βάσει των στοιχείων να μην μπορεί πια να είναι μέλος της ζώνης του ευρώ και να αναγκαστεί να αποσυρθεί από την ζώνη του ευρώ. Δεύτερο ερώτημα. Αν δείτε τι γίνονται σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τι σχεδιάζεται να γίνει σε νομοθετικό επίπεδο για να αντιμετωπίσει κανείς το πρόβλημα των λεγόμενων σκιωδών τραπεζικών φορέων, των εκτός ισολογισμού πιστοτικών φορέων. Θεωρείτε ότι έχετε επιτύχει επαρκή έλεγχο στον τομέα αυτών των ε, ιδρυμάτων εκτός ε, ισολογισμού. Και πολλοί παρατηρητές, το τρίτο ερώτημα είναι, λένε ότι θα πρέπει στη μέση του επομένου ε, έτους θα πρέπει εσείς να δώσετε μια πρόσθετη ρευστότητα της τάξης των 200-400 ε, δισεκατομμύριων ευρώ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κάνετε ή όχι. Στο πρώτο σημείο που θέσατε, ποτέ δεν ανέφερα την Ελλάδα στα εισαγωγικά μου σχόλια. Είχα ένα ερώτημα που αφορούσε την Ελλάδα. Δεν την ανέφερα εγώ ίδιο στην Ελλάδα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η Ισλανδία και η Ελλάδα αναφέρθηκαν σε ένα ερώτημα και εγώ απάντησα στο ερώτημα. Όπω θα έπρεπε και πάντα πρέπει. Ποτέ δεν ανέφερα το όνομα Αργεντινή. Και απαντώντα άλλο ερώτημα για την Ελλάδα, είπε ο ίδιο. Τα σχόλιά μου ισχύουν για οποιαδήποτε χώρα. Οποιαδήποτε χώρα. Και είναι ξεκάθαρο ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και στην περίπτωση της Ιρλανδίας, παραδείγματο χάρη, αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση που είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Στην περίπτωση τη Ιρλανδία, σκληρότατε αποφάσει ελήφθησαν από την κυβέρνηση. Και σωστά. Και σωστά διότι η κατάσταση ήταν δύσκολη και είπα ότι είχα κάθε εμπιστοσύνη ότι παρόμοια θαραλέα και απόλυτα αναγκαία μέτρα, απόλυτα αναγκαίες αποφάσεις θα ληφθούν και στην περίπτωση της Ελλάδας. Αλλά αυτό είναι σχόλιο που ισχύει για όλες τις χώρες. Για όλες τις χώρες ισχύουν αυτά που είπα. Και αληθεύει σε διάφορους βαθμούς σοβαρότητας, όπως βλέπουν όλοι, αλλά αληθεύει ότι αν μπορείς να βασιστείς σε αξιόπιστη στρατηγική μέσω μακροπρόθεσμα, αυτό είναι βασικότατο στοιχείο που σου επιτρέπει να προωθήσεις ανάπτυξη, να προωθήσεις ανάκαμψη. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, αφορούσε τις σκιώδεις τράπεζες. Θα έλεγα ότι αυτό που κάνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, ευρωπαϊκό επίπεδο, και σε επίπεδο της Επιτροπής της Βασιλείας είναι να αποφύγουμε να παγιδευτούμε εκ νέου σε αυτή την ανομαλία των σκιωδών τραπεζών που ήταν βασική γενεσιουργός αιτία για το δράμα που ζούμε όλοι μας και ζήσαμε όλοι μας πρόσφατα. Και επιθυμούμε διακαώς όλη αποφυγή μιας τέτοιας ανομαλίας ένα μεγάλο, ας αφήσουμε εκτός ένα μεγάλο κομμάτι των κινδύνων για τους χρηματοστικούς οργανισμούς που προέκυπτε από μια έλλειψη της ακριβούς αντιλήψης της ενίας Πήραμε διάφορες αποφάσεις. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Eurosystem, η Ευρωπαϊκή Ομάδα θα έλεγα, της Ευρωζώνης πήραμε αποφάσεις όπως όλες οι άλλες κεντρικές τράπεζες στον κόσμο όπως η ομολογή μας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού βρεθήκαμε σε άκρως απαιτητική κατάσταση δύσκολη ανταποκριθήκαμε και νομίζω το κάναμε αυτό γρήγορα ήμασταν τολμηροί όπου χρειαζόταν όμως Δεν χάσαμε την πηξίδα μα. Δηλαδή θέλαμε σταθερότητα τιμών. Αξιοπιστία όσον αφορά σταθερότητα των τιμών. Και άρα είχαμε βάσιμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Εδρεωμένες προσδοκίες πληθωρισμού. Παραμείναμε στα πλαίσια των προσδοκιών για τον πληθωρισμό, των προβλέψεων, κάτω από 2% αλλά κοντά στο 2% με άλλα λόγια. Και όσον αφορά και την λήξη της προσπάθειας που κράτησε ένα χρόνο, όλα όσα κάνουμε σε αυτό το πλαίσιο, τα κάνουμε για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις περιστάσεις όλοι. Να διατηρήσουμε την αξιοπιστία που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αυτό πιστεύουμε όχι μόνο διότι μας ζητούν οι συνάνθρωποι μας να το κάνουμε αυτό και το απαιτούν οι συνθήκες, αλλά και επειδή είναι ένας πολύ αξιόλογος τρόπος να διατηρήσουμε μέσω μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη και ευμάρεια. Και αυτό μας βοήθησε σημαντικά την περίοδο της κρίσης. Διότι αποφύγαμε την υλοποίηση του κινδύνου της, του αποπληθωρισμού. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό τη στιγμή της α, αμέσως μετά την κρίση των Lehman Brothers. Της Lehman Brothers. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Επόμενος είναι ο Σλόβομιρ νίτρα. και σα ζητώ και πάλι να αποφύγετε να θέτετε τρία ερωτήματα τα οποία δεν μπορούν να χωρέσουν σε τρία λεπτά γιατί κάποια μέλη δεν θα προλάβουν να θέσουν τι ερωτήσει του. αν συνεχίσει έτσι κατάσταση ο κ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ δεν θα επαναλάβω τα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί προηγουμένω, παρά το γεγονό ότι πάντα μπορεί κανεί να συμπληρώσει αυτά τα ερωτήματα. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η δική σα αξιολόγηση σε σχέση με το χρονικό ορίζοντα των φορέων εποπτείας που χρειάζεται να δημιουργηθούν. Δεν έχουμε κοινού πιστοτικού θεσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν σημαντικέ διαφορέ <clears throat> μεταξύ των χωρών μα. Υπάρχουν χώρε που έχουν τοπικού φορεί σε ορισμένε αγορέ. Σε άλλε περιπτώσει έχουμε την κυριαρχία μεγάλων διεθνών φορέων κτλ. Βλέπετε λοιπόν να υπάρχει μια απειλή χωρίς να διαμφισβητώ το θέμα της τραπεζικής εποπτείας. Θεωρείτε ότι σε αυτή την πρώτη περίοδο λειτουργία της αυτό το σύστημα εποπτείας με ενδεχόμενη διαμεσολάβηση δεν θα οδηγήσει στον κίνδυνο να αποσταθεροποιηθούν οι τοπικές αγορές και ιδίω οι αγορές αυτές όπου κυριαρχούν μεγάλοι πιστοτικοί φορείς οι οποίοι έχουν την έδρα τους εκτός της ε, χώρας στην οποία δρούν. Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα αυτό. Μια πρώτη παρατήρηση. Πιστεύω ότι όταν εξετάζουμε την πραγματικότητα και την κατάσταση σε όλες τις χώρες που δεν είναι στην ζώνη του ευρώ και είναι παρόλα αυτά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γεγονός όπω το δείχνει και το ερώτημά σα, ένα μεγάλο μέρος του τραπεζικού τομέα έχει να αντιμετωπίσει την παρουσία ξένων πιστοτικών φορέων και αυτό διαδραμάτισε ένα ρόλο ο οποίος ήταν τελικά, αν μπορώ να το πω, σταθεροποιητικού χαρακτήρα. Γιατί αυτές οι τράπεζες είχαν πράγματι τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν ρευστότητα από τον γενικότερο όμιλό τους, από τη μητρική εταιρεία κτλ. Όταν εντατικοποιήθηκε η κρίση και εμείς εστιάσαμε σε αυτά τα έκτακτα όχι στάνταρ μέτρα τα οποία λάβαμε, είπαμε στις τράπεζες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εφόσον έχετε θηγατρικές εταιρείες στην κεντροανατολική Ευρώπη εκτός της ζώνης ευρώ θα πρέπει να συνεχίσετε να παρέχετε ρευστότητα στις τράπεζες αυτές. Μας ενδιέφερε η σταθερότητα όλου του τραπεζικού φορέα, το τομέα μάλλον στην Ευρώπη και είπαμε σε αυτές τις εταιρείες ότι έχετε ευθύνη ως όμιλη τραπεζική και επιστοτική και για τις θηγατρικές σας στην κεντροανατολική Ευρώπη. Αυτό ήταν το τμήμα του μηνύματος το οποίο τους δώσαμε τότε και το οποίο τους θέλουμε τώρα. Σε ό,τι αφορά τώρα τον αντίκτυπο των νέων αυτών αρχών και πάλι, όπως ελέγχθη, όλα εξαρτώνται για την χρονική αλλουχία των γεγονότων από την απόφαση του Κοινοβουλίου. Τώρα σε ό,τι αφορά την επιρροή που μπορούσαν να έχουν αυτοί οι νέοι φορείς, εγώ δεν με τον φόβο αυτό που υποβόσκει στο ερώτημά σας. Νομίζω ότι έχει υπάρξει η απαιτούμενη ισορροπία δεν βλέπω λοιπόν να υπάρχει από χρόνο λόγος να φοβόσαστε μια αθέμητη κατά κάποιο τρόπο λειτουργία αυτών των φορέων όταν έχουν να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα προβλήματα στη χώρα σας. Κύριος Λάγκεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να τονίσω και πάλι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα έδρασε σε αυτή την κρίση με πολύ γαλήνιο και σόφρονα τρόπο και ένα μεγάλο μέρος της σταθεροποίησης οφείλεται στη δική σας δράση. Για τους συστημικούς τώρα κινδύνους. Έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ οι χρηματαγορές. Έχουν περάσει από το να είναι τρεις φορές μεγαλύτερες από την πραγματική οικονομία στο ενδεκαπλάσιο πια το 2007. Μήπως πρέπει να μειωθεί η έκταση των χρηματαγορών και να ξαναγυρίσουμε στο επίπεδο του 2000, δηλαδή τρεις φορές μονάχα. Και τι έχετε να πείτε σε σχέση με την πρόταση των ε, Αμερικανών να αντιμετωπίσουν τα θέματα της διασύνθεσης μεταξύ των τραπεζών που οδήγησε στο να γίνουν κάποιες τράπεζες ακόμα μεγαλύτερες από ό,τι ήταν στο παρελθόν και όχι μικρότερες μέσα στο συστημικό κίνδυνο. Μήπως θα πρέπει να λάβουμε την ε, υπόψη και την ανάγκη να υπάρχει διαφάνεια σε ό,τι αφορά τους ισολογισμούς των πιστοτικών ε, ιδρυμάτων, γιατί ένα μέρος του προβλήματος και που οδήγησε στην κρίση είναι ότι δεν αντανακλώνται όλοι οι κίνδυνοι στον ισολογισμό της. Και επίσης το θέμα ότι πολλές φορές οι τράπεζες δεν ε, αξιολογούν και δεν χρησιμοποιούν την ρευστότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημά σας και ευχαριστώ πολύ και για την πρώτη σας παρατήρηση. Όσον αφορά το συστημικό κίνδυνο, με ρωτήσατε εάν η συρρήκνωση των ε, χρηματοπιστωτικών αγορών, του τραπεζικού τομέα, γενικώ του χρηματοπιστωτικού τομέα, με ρωτήσετε αν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, δεν είναι πολύ εύκολη η απάντηση. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε από όλες τις πλευρές. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε στο ECRB είναι να δούμε το κίνδυνο αυτόν, το συστημικό, ε, υπό το φως αυτής της πολύ κακής εμπειρίας. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη πολλά φαινόμενα. Ήθελα λοιπόν να πω το εξή. Επειδή είπατε και εσεί, αναφερθήκατε στην κατάσταση, ε, στη διαφορά ανάμεσα στο 2000 και το 2007, κατάσταση των παραγόγων. Είπατε ότι έχει πολλαπλασιαστεί ε, σε μία περίοδο 7-8 ετών. Είναι πράγματι ε, περίεργο αυτό. Είναι περίεργο τι είδους φαινόμενο μπορεί να είναι ο λόγος μιας τέτοιας ε, αλλαγής, ενός τέτοιου πολλαπλασιασμού είναι μια ραγδαία εξέλιξη την οποία πρέπει κάπως να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει λοιπόν να τεθεί αυτό το ζήτημα. Και μάλιστα με συστηματικό τρόπο. Και ελπίζω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο τέτοιου είδους ζητήματα πρέπει να τίθενται και σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών και γενικότερα σε επίπεδο ε, παγκόσμιας οικονομίας ε, όταν γίνεται διάλογος. Θα έλεγα και το ίδιο για ε, τα κεφάλαια. Ε, υπήρξε το ίδιο πρόβλημα και ο πολλαπλασιασμός ήταν επί έξι αυτή τη φορά. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτό είναι ή όχι ένας παράγων ε, σταθερότητας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Αλλά θα ήθελα να επαναλάβω ότι δεν θα έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι στην ε, ε, αντιμετώπιση μας. Δεν πρέπει να αντιδράσουμε πάρα πολύ ενθερμό. Πρέπει πραγματικά να το εξετάσουμε σε όλες του τις λεπτομέρειες υπάρχουν, ε, υπάρχει και το θέμα βέβαια της ε, αύξησης της οικονομικής ε, δραστηριότητας όπως είπατε και εσείς ό,τι για να κάνουμε όμως δηλαδή είτε πούμε α, είναι πάρα πολύ, έχει ξεφύγει η κατάσταση είναι πολύ ψηλά τα επίπεδα αυτή είναι μια πολύ απλοϊκή ε, εκτίμηση της κατάστασης, ε, αν είναι πάρα πολύ μεγάλη η διασύνδεση του τραπεζικού συστήματος, είναι κάτι το οποίο πραγματικά χρήζει περαιτέρω ε, ανάλυσης, αλλά πραγματικά στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Αν η δική μου εκτίμηση είναι ότι πρώτα πρέπει να δούμε τη διασύνδεση όλων των φορέων για να μπορέσουμε να να αξιολογήσουμε τον πραγματικό συστημικό κίνδυνο και αν χρειάζεται να αυξήσουμε τη δραστηριότητά τους γιατί πρέπει καταρχάς να δούμε τι είδους κίνδυνος υπάρχει και δεύτερον παρά το γεγονός ότι θα έχουμε προβλέψει μια διαδικασία αντιμετώπισης του κινδύνου σε περίπτωση ε, ε, ε, της κατάρρευσης, υπάρχει πάντοτε μία δυνατότητα βελτίωσης του νεμικού πλαισίου ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για το ίδιο το σύστημα. Και αυτό βέβαια θέλει πολύ σκληρή δουλειά. πρέπει να βελτιώσουμε και την ανθεκτικότητα του συστήματος. Γιατί η συστημική επιρροή του κάθε ιδρύματος ε, μπορεί να εξαρτάται και από το πόσο ευαίσθητο είναι το σύστημα στο σύνολό του. Η Ιλιάνα Ιβανόβα. Ευχαριστώ κύριε Τρισέ που είσαστε εδώ σήμερα μαζί μας. Έχω δύο σύντομες ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση σχετίζεται με τη στατηγική εξόδου και το κόκκινη σημαία, το κόκκινο σημαίακι που αναφέρατε στην αρχή, δηλαδή το σημαδάκι αυτό που είναι οι φορολογικές ανισορροπίες. Πολλές χώρες Ευρωπαϊκή Ενώσης τεράστια χρέη και αυξανόμενα ελλείμματα του προπολογισμού αυτή η απόσυρση της περαιτέρω ρευστότητα, τι συνέπειες θα έχει, ποια θα είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς υπερχρεωμένες χώρες όταν δεν υπάρχει πλέον τρόπος να υποστηρίξουν τη ρευστότητα και να επικρατούν οι πρώτερες ευνοϊκές συνθήκες. Δεύτερο ερώτημα αφορά τα κράτη-μέλη που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι χώρε Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενθαρρύνουν τη διαδικασία οικονομική και νομοσμετική ολοκλήρωση και διεύρυνση της Ευρωζώνης, κυρίως στα πλαίσια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσεως. Ερώτημα. Πώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη, ούτως ώστε αυτές να μπουν στην Ευρωζώνη, κυρίως όταν έχουμε αποδείξει ιστορικό καλής δημοσιονομικής πειθαρχίας, φορολογικής πειθαρχίας. Πώς θα δείξετε σε αυτές τις χώρες ότι ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση. Απάντηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το πρώτο ερώτημα. Έχουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακολουθείτε βιώσιμη στρατηγική όσον αφορά τη φορολογική πολιτική μέσω και μακροπρόθεσμα. Επίσης, με χαρά μου λέγω, ότι αυτό το συνέστημα, αυτή η άποψη είναι κάτι που υποστηρίζει η ECOFIN και η Eurogroup. Και λήφθησαν πολλές αποφάσεις στην τελευταία συνεδρίαση του ECOFIN που ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση. Υποστηρίζουμε απόλυτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ρόλο που διαδραματίζει, που είναι δύσκολος. Αλλά τα πήγε καλά σε άκρως δύσκολες περιστάσεις και υποστηρίζουμε ένθερμα τους δρόμους, τους αυτοκινητοδρόμους που καθόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το αποφάσισε ο εκτελεστικός κλάδος και καλούμε τις χώρες να εφαρμόσουν τα αποφασιστέντα. Και κάποιες χώρες πρέπει να λάβουν τις ενδεδειγμένες αποφάσεις τις επόμενες εβδομάδες. Όσον αφορά τη διεύρυνση της Ευρωζώνης, θεωρούμε ότι είναι κάτι σημαντικότατο, απαιτεί την απαιτούμενη, την δεδειγμένη σύγκληση, κάτι που αναφέρουν οι συνθήκες. Όλες οι κυβερνήσεις θεωρούν σημαντικό το σεβασμό της συνθήκης και πάντα λέγω ότι είναι σημαντικότατο για τις χώρες που εισέρχονται στην Ευρωζώνη να είναι πλήρως έτοιμες. Και αυτό για τη δική τους ευμάρεια, διότι αν δεν είναι απόλυτα έτοιμες, οι χώρες θα αντιμετωπίζουν προβλήματα εντός της Ευρωζώνης. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό και για την Ευρωζώνη. Δηλαδή να συνεχιστεί η παρούσα αξιοπιστία. Το έχουμε υποσχεθεί σε όλους τους λαούς της Ευρωζώνης αυτό. Έτσι βλέπουμε λοιπόν τα πράγματα. Ε, ευχαριστώ για την S&D Λούφινξεν. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τρισέ που ήρθε για να απαντήσει στις ερωτήσεις μας. Όπως γνωρίζετε η ενεργία είναι πολύ υψηλή σε όλη την Ευρώπη και τα επίπεδα, τα ποσοστά απασχόλησης μειώθηκαν κατά πολύ και ακούμε ότι η ανάπτυξη ίσως βελτιωθεί του χρόνου και βλέπουμε ήδη κάποιους τομείς να βελτιώνονται παρόλο που ξεκινάμε από πολύ χαμηλά. Δυστυχώς η ανεργία αυξάνεται και εκείνοι που υποφέρουν περισσότερο συχνά είναι εκείνοι που εργάζονται υπό ασταθείς συνθήκες στην αγορά εργασίας και έχουν χαμηλά επίπεδα κατάρτισης και παιδείας. Υπάρχει ο κίνδυνος να παραμείνει μεγάλη ανεργία. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα τι πιστεύει, πώς μπορεί να μειωθεί η ανεργία, τι είδους οικονομική πολιτική, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για την κατάρτιση Φερρυπίν. Τι πιστεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι θα πρέπει να γίνει. Απάντηση του κ. Τρισέ. Ναι, καταρχάς έχετε απόλυτο δίκιο. Την τρέχουσα περίοδο αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερες δυσκολίες διόλου των συνεπειών υστέρηση, χρονική υστέρηση. Η ύφεση δημιούργησε πολλές δυνατότητες αυξήσεω της ανεργία και βλέπουμε η ανεργία πράγματι να αυξάνεται ακόμα και αν Τώρα μπαίνουμε στα μαύρα στοιχεία, μπαίνουμε στα θετικά στοιχεία. Δεν αρκούν όμως αυτά για να αντισταθμίσουν τις συνέπειες που έρχονται με καθυστέρηση από την προηγηθήσα ύφεση. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι κακό για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και γι' αυτό επιμένουμε και προωθούμε όλα τα μέτρα που μπορούν να αυξήσουν την εμπιστοσύνη και θα μπορέσουν να επιτρέψουν στην ευρωπαϊκή οικονομία και την οικονομία της Ευρωζώνης και της Ευρώπης γενικά να ωφεληθεί από, το, τη βελτίωση της εμπιστοσύνης. Όσον αφορά την απασχόληση, σαν βασική αρχή θεωρούμε ότι οι διαθροτικές μεταρρυθμίσεις που αποφασίστηκαν από την Ευρώπη, από όλους τους εκτελεστικούς κλάδους, θα επέτρεπαν μια πιο ενεργή, πιο δυναμική οικονομία που θα δημιουργούσε και περισσότερες θέσεις απασχόλησης αν όλα πήγαιναν καλά. Αυτό ισχύει για όλα τα θέματα της ατζέντα της Λισαβόνας που αποφάσισαν όλες οι κυβερνήσεις. Θεωρούμε ότι εντός του προγράμματος της Λισαβόνας Εντό των δομικών μεταρρυθμίσεων που ενδείκνυνται και υποδεικνύονται, μεταρρύθμιση τη εκπαίδευση και τη κατάρτιση έχει εξαιρετική σημασία. Είμαστε στην τεχνολογία τη γνώση και όλο και θα αυξάνεται αυτή, θα επικρατεί περισσότερο η οικονομία τη γνώση. Και ο επιμερισμό τη αγορά εργασία, μάλλον η αγορά εργασια θα χαρακτηρίζεται περισσότερο από την ανάγκη για ανθρώπου που γνωρίζουν την αγορά της γνώση θα, θα θέλουμε περισσότερα εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες που θα δίνουν μεγάλη προστιθέμενη αξία και υπηρεσίες και αγαθά που θα βασίζονται σε αυξημένη, σε προθυμένη τεχνολογία. Χρειάζεται προσπάθειες εκεί. Πιστεύουμε ότι σε αρκετές χώρες θα πρέπει να γίνουν και όσον αφορά την αγορά εργασίας δομικές αλλαγές είναι πάρα πολύ σημαντικές για να προωθήσουν την ε, ανάκαμψη και την, ανάκαμψη και την οικονομική ε, ανάπτυξη και να δημιουργήσουν τις απασχόλησεις. Πίτερ Σίμων. Κύριε Πρόεδρε, εμείς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση και να αποτρέψουμε μελλοντικές ε, κρίσεις. Έχετε εξασφαλίσει ότι ξέρουμε πώς έχουμε καταλήξει αυτή την κρίση και πώς απέτυχε το σύστημα το χρηματοοικονομικό. Ο κύριος Άκερμαν, ο πρόεδρος της ε, Deutsche Bank, έκανε μια πρόταση προς την ε, κοινή γνώμη και είπε ότι ήδη από τώρα θα πρέπει ο τραπεζικός κόσμος αλλά και ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να κάνουν κάποιες εξοικονομήσεις να δημιουργήσουν ένα μαξιλάρι, ένα αποθεματικό για την περίπτωση που ξεσπάσει και μια νέα κρίση. Αυτό οδήγησε σε κάποια οργή και αγανάκτηση στην κοινή γνώμη της ε, Γερμανίας που δεν μπορούν να δεχτούν ότι, ότι οργανισμοί όπως η Deutsche Bank που έχουν σαν στόχο την ταχεία κερδοφορία θέλουν να κοινωνικοποιήσουν τις, ήδη, τις που ήδη υπέστησαν. Θα ήθελα να έχω την άποψή σας σε σχέση με μια τέτοια προσέγγιση. Πρώτα απ' όλα <clears throat> είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι το σύνολο σύστημα, το σύνολο χρηματοοικονομικό σύστημα θα είναι ανθεκτικό. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε ό,τι αφορά την εποπτεία. Ο στόχος μας φυσικά είναι με τον απόλυτο σεβασμό για τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν θα πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας αλλά σίγουρα θεωρούμε ότι ήδη από το 2012 οι, κεφαλουγικές, οι απαιτήσει κεφαλουγικής επάρκειας θα πρέπει να είναι σημαντικότερες από ό,τι είναι τώρα, ώστε όλα τα πιστοτικά ιδρύματα μεμονωμένα να είναι πιο ανθεκτικά, επομένως και το σύστημα να είναι πιο ανθεκτικό. <clears throat> Επομένως, η ιδέα αυτή του να δημιουργηθούν αποθεματικά, αυτό είναι καλό να έχουμε αποθεματικά για να αντιμετωπίσουμε δύσκολες στιγμές. Αυτό είναι μια λογική αντιμετώπιση. Προβλέπουμε επίσης να έχουμε μέτρα τα οποία θα είναι αντικυκλικού χαρακτήρα, θα κινούνται αντίθετα με τον οικονομικό κύκλο και θα επιτρέψουν μέσα στο πλαίσιο της ε, Βασιλείας 2 σε συστημικό επίπεδο κάθε συγκεκριμένος πιστοτικός φορέας να δημιουργεί ένα αποθεματικό, ένα κατάλληλο αποθεματικό για να μπορέσει να αντιμετωπίσει δύσκολες περιστάσεις στο μέλλον. Τώρα το να ζητήσουμε από τις κυβερνήσεις εκ των προτέρων να συσσωρεύσουν ένα αποθεματικό το οποίο ενδεχομένως θα είναι απαραίτητο για να αποτρέψει νέα προβλήματα στο μέλλον αυτό είναι θέμα κυριαρχίας των Εθνικών Κοινοβουλίων κατά την άποψή μου. Η δική μου άποψη αυτή τη στιγμή, η δική μου εντύπωση είναι ότι είναι πολύ απίθανο ο φορολογούμενος για δεύτερη φορά θα αποδεχθεί να υποστεί και νέους κινδύνους και νέες δυσκολίες πέραν αυτών που αντιμετωπίσανε με την τωρινή κρίση. Δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα πρόσφορα ένα τέτοιο μέτρο αυτήν τη συγκεκριμένη στιγμή που βρισκόμαστε. Καταρχήν το σύστημα θα πρέπει να γίνει πιο ισχυρό και πιο ανθεκτικό, προτού ζητήσουμε από του φορολογούμενου να βάλουν ακόμα βαθύτερα το χέρι στην τσέπη. Θα δούμε όμω αν, αφού έχουμε πράξει όλα αυτά τα οποία θέλουμε απαραίτητα, αν αυτά θα βοηθήσουν και τον ιδιωτικό τομέα να είναι πιο ανθεκτικός θα δούμε αν θα υπάρξουν περιπτώσεις στο μέλλον που ο φορολογούμενος θα πρέπει και πάλι να πληρώσει την ύφη. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο εγώ μπορώ να το αποκλείσω, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη προσέγγιση στο πρόβλημα για τη σημερινή στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν χώρες στην Ευρωζώνη που έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν και υπάρχουν και χώρες όπως, η Ισπανία για παράδειγμα όπου η έλλειψη ε, διαρθρωτικών αλλαγών ε, σημαίνει ότι θα συνεχίσει η ύφεση. Ε, στην Ισπανία η αγορά ε, σπιτιών έχει, δεν, δεν έχει παρουσιάσει καμία βελτίωση μία ε, νομισματική πολιτική, ενδεχομένως όμως να είναι επώδυνη σε κάποιες χώρες όπως στην ε, Γαλλία και στη Γερμανία. Αρχίζει να είναι θετικός ο πληθωρισμός και σε άλλες χώρες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία εξακολουθεί να υπάρχει αποπληθ ε, αποπληθωρισμός. Ενδεχομένως λοιπόν η νομισματική πολιτική της Ισπανίας λόγω της κατάστασης αυτής τελικά να είναι πολύ περιοριστική. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει έναν τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής ή θα συνεχίσει με αυτήν την νομισματική πολιτική που έχει ως τώρα ακολουθήσει. Και μία ακόμη ερώτηση για την διαφάνεια. Νομίζω ότι η διαφάνεια ενισχύει την ανεξαρτησία και νομίζω ότι είναι σημαντικό ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δημοσιεύει τα αποτελέσματα των ε, συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ε, κάνει για παράδειγμα η Τράπεζα της Ιαπωνίας. Επίσης, Όσον αφορά τα ενέχειρα, θα ήθελα να μην ε, μιλούμε ε, πλέον ε, σε εθνικό επίπεδο, γιατί σε αυτή την κρίση όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Thank you very ευχαριστώ πολύ για την παρατήρησή σας. Μία πρώτη παρατήρηση. βρισκόμαστε σε οικονομική νομισματική ένωση. Το ε, μήνυμα είναι και προς εσάς και προς ε, όλους τους υπόλοιπους ε, συναδέλφους σας που με ρωτούν για την προσχώρηση στην Ευρωζώνη. Βρισκόμαστε σε μία ζώνη ενιαίου νομίσματος. Ε, το ευρώ είναι ένα. Το ίδιο ισχύει και, για την, ε, και προς την ε, Ασία. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα ευρώ για την Ισπανία και ένα ευρώ για κάποιον άλλον. Ένα ευρώ υπάρχει, ένα επιτόκιο υπάρχει, μία συναλλαγματική ισοτιμία υπάρχει για το ευρώ, για όλους. Και βεβαίως υπάρχει και ένα ε, ίδρυμα που είναι υπεύθυνο ε, για την ε, γενική σταθερότητα των τιμών στην Ευρωζώνη για 16 χώρες και ε, μιλάμε για ένα μέγεθος ε, περίπου ίδιο με των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, κανένας δεν θα έλεγε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε σχεδιάζουν την νομισματική της πολιτική για τη Μασαχουσέτη, για την Καλιφόρνια, για τη Φλόριντα. η νομισματική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών καθορίζεται για το σύνολο της, των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ίδιο ισχύει και για μας. με το ευρώ στην Ευρωζώνη. Άρα, μία ακόμη φορά να πω, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, από τη στιγμή που υπάρχει μία καθορισμένη νομισματική πολιτική υπέρ ε, της ευημερίας 330 εκατομμυρίων ανθρώπων, υπάρχουν βέβαια και κάποιες εθνικές αποφάσεις. Υπάρχουν κάποιες εθνικές αποφάσεις όσον αφορά τη φορολογική πολιτική, όσον αφορά την παρακολούθηση ε, της ε, εθνικής οικονομίας και όπως επίσης και για τις διαρθρωτικές αλλαγές. Τώρα, το τι μπορεί να γίνει σε εθνικό επίπεδο εξακολουθεί να παραμένει σημαντικό. Το να καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι ό,τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο ε, έχει κάποια σημασία. Υπάρχει μία εποπτεία ομοτήμων για να το πω έτσι ε, και αυτό είναι καλό και υπάρχει βέβαια και η εποπτεία των διαρθρωτικών πολιτικών όσον αφορά τη διαφάνεια θα ήθελα να πω ότι Είμαστε η πρώτη κεντρική τράπεζα που δημοσιεύει εισαγωγικό σχόλιο 5-6 σελίδων για να εξηγήσει λεπτομερώς ποια ήταν η λογική του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο πριν από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αλλάξαμε τον τρόπο με τον οποίο ε, αλλάξαμε την έννοια της διαφάνειας, σε πάση περιπτώσει. Ήμασταν οι πρώτοι που κάναμε συνεντεύξεις τύπου αμέσως μετά από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο προκάτοχός μου, Βιμ Ντάιζενμπεργκ, το έκανε αυτό για πρώτη φορά. Και είναι ένας τρόπος να είμαστε όσο το δυνατόν πιο διαφανείς, δηλαδή να απαντάμε αμέσως ε, σε ερωτήσεις, αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πέντε με έξι σελίδες εξηγήσεων ε, για ποια, ποια ήταν η διάγνωσή μα, ποια είναι η λογική μας, τι ακριβώς θα κάνουμε. Πιστεύουμε λοιπόν ότι... Δεν είναι σωστό να αναφέρουμε τις ε, μεμονωμένες ψήφους, όταν υπάρχουν και νομίζω ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη βέβαια ότι είναι 16 κράτη ε, μέλη και ε, κάθε κράτος μέλος πρέπει να υπερασπίζεται την απόφαση που έχει ληφθεί από το ε, Συμβούλιο των Διοικητών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Η έχει το πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε για μένα η στρατηγική εξόδου πρέπει να έχει να αποτελείται από μια σειρά βημάτων με το σωστό χρονισμό που θα μας επιτρέψει να εγκαταλείψουμε αυτά τα έκτακτα μέτρα στον τομέα του προϋπολογισμού και της χρηματοοικονομικής πολιτικής, αλλά απαιτεί και τον κατάλληλο μηχανισμό συντονισμού. Αυτό με φέρνει και πάλι στην σύνδεση μεταξύ της νομισματικής εξόδου και της ε, δημοσιονομικής εξόδου. Θα ήθελα να τα δω αυτά τα πράγματα με μια διαφορετική οπτική γωνία από ό,τι συναδελφή μου. Ξέρουμε ότι είναι επικύλων ο αντίκτυπος <clears throat> της κρίσης στα διάφορα κράτη-μέλη. Κάποιες χώρες θα ανακάμψουν νωρίτερα από τις άλλες. Αυτό οδηγεί σε διαφοροποιημένο χρονισμό σε ό,τι αφορά τη στιγμή της δημοσιονομικής εξόδου. Για ορισμένα κράτη-μέλη, όμως, κατά τη δική μου άποψη, είναι απαραίτητο η νομισματική έξοδο να ακολουθεί τη δημοσιονομική έξοδο για να μην υπάρξει μια παγίδα χρέους όταν πρόκειται να πρέπει να ξεπληρώσουν το δημοσιονομικό τους ε, χρέος με υψηλά επιτόκια. Μέσα στο πλαίσιο αυτό λοιπόν θεωρείται ότι η κατάργηση όλων αυτών των ειδικών μέτρων που θα προβεί σε αυτή την άρση των μέτρων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα <clears throat> στο μέλλον να μην οδηγήσει, να μην δώσει λαβή σε αύξηση των επιτοκίων. Γιατί αν υπάρξει η αύξηση των επιτοκίων, αυτό θα υπονομεύσει την ανάκαμψη στην ε, ζώνη του ευρώ. Το επόμενο ερώτημα Θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να αναπτύξει ένα σχέδιο για να εξασφαλίσει το συντονισμό των στρατηγικών δημοσιονομικής εξόδου, ώστε η νομισματική έξοδο στη συνέχεια μπορεί να γίνει στη συνέχεια με τον πιο ομαλό τρόπο που είναι δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο. Ποιο θα ήταν για εσά λοιπόν το θεσμικό πλαίσιο για να υπάρξει αυτή η απαραίτητη μορφή συντονισμού για, τον, για την δημοσιονομική έξοδο, γιατί και η νομισματική έξοδος από την κρίση θα εξαρτάται από αυτή την πρώτερη ε, συντονιστική ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ κυρία. Κυρία μου, έχω να κάνω ορισμένε παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, όπως είπατε και εσείς η ίδια, δεν υπάρχει μια ενιαία αντίληψη δημοσιονομικής εξόδου. Κάποιες χώρες έχουν διαχειριστεί με υποδειγματικό τρόπο την κρίση. Για τις χώρες αυτές λοιπόν το πρόβλημα ουσιαστικά δεν υφίσταται. Άλλες χώρες έχουν υπερχρεωθεί σαν αποτέλεσμα της κρίσης. Κάποιες χώρες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία της δημοσιονομικής εξόδου, παραγωγός χάρη η Ιρλανδία. Άλλες χώρες θα ξεκινήσουν το 2011. Κάποιες χώρες θα ξεκινήσουν το 10, άλλες το 2011. Επομένως αυτή η διαδικασία της εξόδου έχει ξεκινήσει, τουλάχιστον έχει τύχει απόφαση με πρόταση της Κομισιόν να υπάρξει το σύνολο των καταλήλων πολιτικών σε επίπεδο κυβερνήσεων. Δηλαδή αυτό αφορά τη λεγόμενη δημοσιονομική έξοδο από την κρίση. Σε ό,τι αφορά τώρα την υποστήριξη προς τον χρηματοοικονομικό τομέα, την νομισματική έξοδο. Εκεί έχει ξεκινήσει η διέξοδος, η σημαντική αυτή υποστήριξη προς τον χρηματοοικονομικό χώρο που δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότηση των τραπεζών και μέσω και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Δεν έχει καμία σχέση λοιπόν με τις δημοσιονομικές προσπάθειες. Όλα αυτά έχουν σχεδιαστεί όπως και τα μη στάνταρ μέτρα μας για να αντιμετωπίσουν μια έκτατη κατάσταση η οποία εμπόδιζε την ομαλή λειτουργία των χρηματοοικονομικών αγορών αλλά αυτό έχει ήδη ε, ξεπεραστεί σε κάποιο σημείο και όσο βελτιώνονται οι αγορές τόσο και τα έκτακτα αυτά μέτρα χάνουν το ρολό ύπαρξής τους. Εμείς, όπως σας είπα, χρησιμοποίησαμε και συμβατικά και μη συμβατικά <clears throat> μέτρα. Την προηγούμενη Πέμπτη και το τόνισε αυτό ε, θεωρήσαμε ότι τα τωρινά επίπεδα επιτοκίων είναι τα πρέποντα για την τωρινή κατάσταση και το γεγονός ότι εμείς αρχίζουμε την άρση μιας σειράς μη συμβατικών μέτρων δεν έχει αντίκτυπο σε ό,τι αφορά τα επιτόκια. Αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι τα επιτόκια μπορούν να παραμείνουν σε αυτό το σημερινό επίπεδο και δεν έχουμε καμία πρόθεση να περάσουμε κάποιο μήνυμα το οποίο αφορά το επίπεδο των επιτόκιων αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε όλοι ότι έχουμε μόνο μία ένα μπούσουλα, ουσιαστικά μία πορεία πλεύσης. Αν υπάρξει ανάγκη για να διατηρήσουμε τη σταθερότητα των τιμών και η αξιόπιση σταθερότητα των τιμών να τροποποιήσουμε τα επιτόκια, να το πράξουμε εν καιρό. Κυρία Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που αναφερθήκατε στην εισαγωγική σας παρέμβαση για την κεντροανατολική Ευρώπη και την ανάγκη να υπάρξει μια σταθεροποίηση στις χώρες της ε, κεντροανατολικής Ευρώπης. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό γιατί εξακολουθεί να μαστίζεται αυτή η περιοχή από σημαντικά οικονομικά προβλήματα. Πριν από τρία-τρεις μήνες σας είχα θέσει το ερώτημα πώς θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε μέτρα ανταλλαγής swap μεταξύ χωρών της ζώνης του ευρώ και χωρών εκτός της ε, ζώνης του ευρώ. Αυτό δεν έγινε πραγματικότητα απόλυτα. Αν εξετάσουμε όμως την κατάσταση τώρα στην Ουγγαρία. Οι φορείς της αγοράς λένε και παραπονούνται ότι δεν υπάρχει επαρκής ρευστότητα. Είσαστε εσείς ικανοποιημένος με το επίπεδο της ρευστότητας στην ε, Ουγγαρία. Και οι τράπεζες επίσης διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι τα μέτρα για την ε, επανακεφαλαιοποίηση έχουν αρθεί στην ε, ζώνη της Ευρώπης ενώ οι τράπεζες στις χώρες λένε ότι οι χώρες της ζώνη του ευρώ πήραν μια σημαντική, σημαντική ένεση ρευστότητος, αλλά όχι οι χώρες της ε, Ανατολικής Ευρώπης. Επομένως, οι χώρες της ε, ζώνης του ευρώ μπορούν τώρα να ικανοποιούν τις ε, απαιτήσεις κεφαλαιοχικής επάρχειας, αλλά όχι οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Θυμάμαι το ερώτημα που είχα θέσει την προηγούμενη φορά. Να πω μόνο ότι όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Ουγγρική Κεντρική Τράπεζα είναι πολύ στενή σχέση. Σχέση εμπιστοσύνης. Και έχουμε οικονομικές σχέσεις που πρέπει να πω πάνε πολύ καλά. Σχέση μεταξύ των δύο κεντρικών τραπεζών. Θεωρώ μάλιστα ότι αυτό που κάνουμε σαν άμεση συνεργασία με την Ουγγρική Κεντρική Κεντρική Τράπεζα και τα μηνύματα που στέλνουμε στις κεντρικές, ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες, εμπορικές τράπεζες της Ευρωζώνης όταν συνεργάζονται με τους ομολόγους στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είναι διτός. Με δύο τρόπους προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Αυτό που μετράει όμως είναι σαφήνεια της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της ίδιας της χώρας. Αυτό είναι θεμελιώδους σημασίας και βοήθησε σημαντικά. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Τελευταίο ερώτημα. Η Βίκη Φόρτ, Διότι θα πρέπει να πάμε και στον Υπουργό και ε, θέλουμε και χρόνο για το Eye. Ευχαριστώ κύριε Τρισέ. Σαφέστατες οι εξηγήσεις που δώσατε σχετικά με τα όσα πράττει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να βγούμε από την χρηματοπιστωτική κρίση και για τα όσα θα κάνετε με το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Όμω επικρατεί σύγχυση στον εγκέφαλό μου από αυτά που άκουσα. Στην τελευταία συνεδρίασή μα το Σεπτέμβριο συναντήσαμε το ενδεχόμενο συγκρούσεως συμφερόντων, διότι είστε επικεφαλής και των δύο αυτών φορέων και μας είπατε ότι για να παραμείνουν ξεχωριστά τα δύο καθήκοντά σας, όχι μόνο θα υπάρχει ξεχωριστό προσωπικό, αλλά θα είστε υπόλογος και στο Κοινοβούλιο δύο φορές όσον αφορά τον κάθε ρόλο σας. Όμως υπάρχει κάποια διάχυση ευθυνών Και έτσι καταλαβαίνω από αυτά που μας είπατε ότι ίσως δεν έχετε πλέον ξεχωριστούς αυτούς τους ρόλους. Ο έλεγχος. Και, αυτού του ρόλου και των εποπτικών αρχών δεν είναι σαφής. Ευθύνες των φορέων. Ο Ερμάν ανέφερε την Ισπανία. Και πήγε μια αντιπροσωπή τη Επιτροπή μα την περασμένη εβδομάδα στην Ισπανία. Και ναι, υπάρχει μια βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση. Όμως η χρηματοπιστική κρίση απεθέυθη κατά πολύ λόγω πιο πολλής πιο προσεκτική, μάλλον εθνικής ρυθμιστικής προσέγγισης. Η Τράπεζα τη Ισπανίας είχε 70 ανθρώπου στην Τράπεζα Banco Santander ε, για να ρυθμίζουν τα τεκτενόμενα. Η ΣΥΖΑ έχει μέλη του προσωπικού που πάει να τα αυξήσει στους 80. Και FSA στο Λονδίνο έχει 3.000 μέλη. Αυτοί είναι οι φορείς. Ποιες ευθύνες πρέπει να έχουν, πόσες ευθύνες. Όταν είμαι στην τράπεζα, η τράπεζα της Ισπανίας, η τράπεζα της Ισπανίας, οι μεγαλύτερες, οι μικρότερες, οι ρυθμιστικές αρχές, οι εκπρόσωποι των ασφαλιστικών εταιριών, όλοι είπαν ότι η ευθύνη για υποπτία και λήψη αποφάσεων για διάφορε επιχειρήσει θα πρέπει να παραμείνει σε εθνικό επίπεδο, εθνική αρμοδιότης. Εν κατακλείδη το ερώτημά μου είναι συμφωνείτε με αυτά που είπα. Ευχαριστώ κυρία μου, λέει ο κ. Τρισέ. Πρώτα απ' όλα, ε, εάν επιτρέπετε να σας πω ότι είμαι μπροστά σας σαν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν υπάρχει πρόεδρος ε, του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, διότι δεν έχει δημιουργηθεί. Και επιβεβαιώνω απόλυτα αυτά που είπα. Εάν οι συνάδελφοί μου έχουν την καλοσύνη να με διορίσουν σαν πρόεδρο του ESRB, του Συμβούλιου Συστημικού Κινδύνου και βεβαίως θα αναφέρω τα σχετικά με αυτό το Συμβούλιο σε εσά και θα είναι διαφορετική αυτή η παρουσία μου σε σχέση με την παρουσία μου εδώ στον Πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συμβάλλει στη δημιουργία του Συμβουλίου για την Ανάλυση του Κινδύνου, θα δίνει ε, ε, υποστήριξη οικονομική και επιμελητία, όπω αποφασίστηκε. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δει ακριβώς τι θέλει, αλλά επιβεβαιώνω αυτά που είπα. Και είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι δύο διαφορετικές ευθύνε. Είναι απόλυτα ξεκάθαρο αυτό. Όσον αφορά τη θέση της μικροεποπτείας, εν αντιθέσει με την μακροεποπτεία, καταρχάς εκτιμώ τα μάλα το ότι είπατε ότι Καλό είναι η Κεντρική Τράπεζα να συμμετέχει κατά πολύ στην εποπτεία των τραπεζών. Όπως ξέρετε δεν το πιστεύουν αυτό ως ενδεδειγμένο σε όλη την Ευρώπη, αλλά πιστεύουμε ότι ενδείκνυται εμείς και το είπαμε προκαιρού από παλιά. Δεύτερον, βεβαίως όταν έχεις αντιμετωπίσει αντιμετωπίσεις διασυνοριακούς θεσμούς, έχεις πρόβλημα. Ποια είναι η σωστή ερμηνεία της εποπτείας για τον όμιλο εν γέννη. Ε, εξού και η χρησιμότης των αρμόδιων φορέων να κινούνται καταλήλως. Γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν σημαντικό σε αυτή την περίπτωση να έχουμε πανευρωπαϊκή επισκόπηση όσον αφορά την μικροεποπτεία υπό την προϋπόθεση ότι έχεις απέναντί σου υπερεθνικούς θεσμούς, πολυεθνικούς θεσμούς και όχι έναν εθνικό, ένα εθνικό φορέα. Συμφωνώ μαζί σας. Όμως υπάρχει ανάγκη γενίκευσης γενικής χρήσεως των αρχών και των ενιών που θεωρούνται καλές. Και ισπανικός εποπτικός φορέας δυναμικά εισήγαγε μια αρχή που δεν χρησιμοποιείται γενικά στα πλαίσια της Επιτροπής της Βασιλείας και της Ευρώπης ή σε παγκόσμιο επίπεδο. Όμως η αρχή αυτή απεδείχθη άκρως χρήσιμη υπό τις περιστάσεις αυτές. Η ιδέα λοιπόν σε επίπεδο ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, αν θέλουμε μια τέτοια ενιαία αγορά, με αποφασιστικότητα το ίδιου κανόνες για την εποπτεία τραπεζών εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ φυσικό και πιστεύω ότι προ τα εκεί κινούμεθα. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται μια κεντρική αρχή, ένας κεντρικός φορέας για να κάνει τις απαραίτητε διευθετήσεις σε περίπτωση διαφωνιών που ελπίζω να μην συμβαίνει συχνά μεταξύ των διαφόρων φορέων μικροεποπτείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω στην επόμενη φορά που θα ξανάρθει ο κύριος Τρισένα να ε, γνωρίζουν ότι ε, θα πρέπει να κάνουν ε, δύο ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουν όλα καταγραφεί, όλα όσα μας είπατε και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σε τρεις μήνες. Δεν ξέρω ακριβώς πότε όμως, δεν έχω ημερομηνία. Ευχαριστώ πολύ. Okay, can you take your seats again now that the minister is with us? Καθίστε παρακαλώ, γιατί ήρθε ο Υπουργός. Colleagues, can you, can you take your seats? Μπορείτε να καθίσετε παρακαλώ. Για να ακούσετε και τον Υπουργό. Είναι εδώ υπουργός ε, της ε, Προεδρίας, που σύντομα θα είναι απερχόμενη, να μας πει ορισμένα πράγματα για το τι συνέβη, τι περιμένει την επόμενη Προεδρία και μετά με τη διαδικασία ΚΑΤΣΙΑΙ θα ακούσουμε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι εδώ και ώστε να μπορώ να σας πω τι ε, καταφέραμε στα συμβούλια ΕΚΟΦΗΝ κατά τους τελευταίους έξι μήνες. Αυτοί οι έξι μήνες ε, Βέβαια ήταν ε, μια πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περάσαμε τη χειρότερη και την πιο προβληματική περίοδο ε, στο ΑΕΠ ε, παρατηρήθηκε πτώση τουλάχιστον 5% και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κατά πάσα πιθανότητα θα χάσουμε ακόμη 4% συνολικά. Η ανεργία αυξάνεται, έχει ήδη φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα σε πολλές χώρες και κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει να αυξάνεται το 2010 και ενδεχομένως και πιο μετά. Τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί κατά τον τελευταίο χρόνο για την αντιμετώπιση της κρίσης ε, ήταν ε, ιδιαίτερου φάσματος ε, και προς όλες τις κατευθύνσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε με ενισχυμένη συνεργασία να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό τομέα και γενικότερα στην οικονομία. Υπήρξαν συγκεκριμένα προγράμματα εγγυήσεων ε, προ τη της ε, σταθεροποίησης των ε, χρηματοπιστωτικών αγορών και υπήρξε και συντονισμό όσον αφορά τι οικονομικές πολιτικέ στο πλαίσιο του προγράμματο οικονομικής ανάκτηση που προσπάθησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να σταθεροποιήσει την κατάσταση. Τώρα, Όσον αφορά την ε, Σουηδική Προεδρία αυτή καθεαυτή, επικεντρωθήκαμε κυρίως ε, σε τέσσερις τομείς. Ο ένας τομέας είναι καταρχάς ε, η υποδομή των χρηματοπιστωτικών αγορών, η αποφάσει όσον αφορά την, τις νομές εποπτείας, όπως επίσης και τις οδηγίες για τις απαιτήσει σε κεφάλαια και τη διαχείριση κινδύνου, τη βελτίωση της διαχείρισης κινδύνου που σκοπό είχε να διευκολύνει τη στρατηγική εξόδου από τα έκτακτα μέτρα. Η δεύτερη προσπάθεια αφορούσε τα δημοσιονομικά μέτρα που ελήφθησαν ε, επειδή υπήρχε πολύ μεγάλο έλλειμμα. και σχετική απόφαση στην, στο τελευταίο Συμβούλιο. Κάτι ακόμη ε, που μας απασχόλησε είναι το θέμα του κλίματος. Αρχίζει σήμερα η Σύνοδος στην Κοπενχάγη ε, η χρηματοδότηση της ε, κλιματικής αλλαγής ήταν ένα σημαντικό θέμα του προγράμμα, ένα σημαντικό, μια σημαντική προτεραιότητα του προγράμματός μας. Ε, επίσης επικεντρωθήκαμε και πάρα πολύ στον συντονισμό της θέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του G20 και βέβαια ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους καταλήξαμε στην πολύ δύσκολη κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή είναι βέβαια η έλλειψη ε, ε ρυθμιστικών ε, κανόνων, ότι υπήρχαν φοβές, δηλαδή αδυναμίες ε, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους σοβαρές κρίσεις. Συνεπώς και για την μακρό και για την μικρό εποπτεία, Έγιναν σημαντικέ προσπάθειε κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα. Στην τελευταία συνεδρίαση του ΕΚΟΦΗΝ την περασμένη εβδομάδα καταλήξαμε σε μια συμφωνία να λάβουμε μια απόφαση ε, για έναρξη συζητήσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την μακροεποπτεία. Είχαμε ήδη λάβει στο παρελθόν αποφάσει όσον αφορά ε, ε, το θέμα αυτό και νομίζω ότι ο βαθμός συνεργασίας όλων των κρατών μελών στο Συμβούλιο ήταν ε, αρκετά υψηλός. Ε, τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη ήθελαν να πάνε κάπως παραπέρα για να ε, καταλήξουμε σε κάποια απόφαση. Τώρα, όσον αφορά το νέο Συμβούλιο Αξιολόγησης του Συστημικού Κινδύνου, θα είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του για τη βελτίωση της ε, δυνατότητας αξιολόγησης των ε, κινδύνων και επίσης θα επικεντρωθεί ε, στο θέμα της οικονομικής αστάθειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την πιο μακροπρόθεσμη σταθερότητα και βιωσιμότητα. Όσον αφορά τώρα την μακροπιστωτική εποπτεία, που είναι νομίζω και αυτό ένα σημαντικό επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που, για το οποίο πρέπει να ε, επενέσουμε τον κύριο Ντελαροζιέρη, είναι ότι δεν επέλεξε την ε, καλύτερη λύση, αλλά την εφικτή λύση. Καταφέραμε, συνεπώς, να καταλήξουμε σε ένα σύστημα που βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές, οι οποίες όμως δεν θα είναι τέλειες για κάθε κατάσταση, αλλά μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα, για να μπορέσουν, τα ζητήματα που μας εμποδίζουν να έχουμε μια μακροπιστωτική σταθερότητα. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν εξαιρετική η δουλειά και, η Επιτροπή, και της Επιτροπής Δελαροζιέρ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ήταν πολύ καλή. Ε, τέθηκαν τα θεμέλια για καλύτερη ε, ρυθμιστική δομή και επίσης όσον αφορά τις ε, μακροοικονομικές στατιστικές νομίζω ότι ήταν πολύ καλά τα αποτελέσματα της προσπάθειας που υπήρξε ε, και με τη νέα ομάδα που συστάθηκε αλλά και στο πλαίσιο του συντονισμού των κρατών μελών και νομίζω ότι η δραματική εμπειρία του περασμένου φθυροπόρου ήταν αυτή που μας όφησε να βρούμε μία λύση. Και επίσης υπήρξε και πρόοδος σε σχέση με την άποψη που είχαν ορισμένα κράτη-μέλη για την εθνική προσέγγιση τέτοιου είδους ε, κρίσεων και ειδικότερα όταν για συνοριακή φύσεω. Επίση, ε, υπήρξε και ένα συμπέρασμα του Συμβουλίου όσον αφορά την στρατηγική εξόδου είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τα μέτρα αυτά για κάποιο χρονικό διάστημα, γιατί είναι σημαντικό να σταθεροποιηθεί ο χρηματοπιστωτικό τομέα για ε, κάποιο ε, χρονικό διάστημα ακόμη, αλλά είναι επίσης ε, προφανές ότι πρέπει σιγά να αρχίσουμε να αποσύρουμε ορισμένα τέτοια μέτρα και χρειάζεται μια συντονισμένη στρατηγική για να γίνει αυτό, γιατί υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν συνέπειες και σε άλλες πολιτικές, αλλά και συνέπειες και στην ανταγωνιστικότητα ε, των κρατών μελών. Κάτι ακόμη για την χρηματοπιστωτική υποδομή είναι το θέμα της οδηγίας απαιτήσει ε, σε κεφάλαια CRD3 ο βαθμός της κεφαλαιοποίησης των τραπεζών, όπως επίσης και η ικανότητά τους ε, να διαθέτουν κεφάλαια για να μπορούν να αντιμετωπίσουν ε, ε, καταστάσεις κρίσεων. Κάτι το οποίο θα βοηθήσει τον τραπεζικό τομέα και μακροπρόθεσμα. Τώρα, όσον αφορά τις μεγάλες συζητήσεις για τα μπόνους, Προφανώς αυτό ήταν ένα μεγάλο τμήμα τη προπαρασκευαστικής εργασίας για την ε, ομάδα G20 και οι αρχές που αναφέρονται στην οδηγία περί απαιτήσεων ε, κεφαλαίων είναι ότι θα υπάρξει μία αναστολή των πληρωμών των πόνους ώστε να υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του κέρδους αλλά και τη μακροπρόθεσμη σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Βέβαια είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μα απασχολήσει ξανά. Είναι προφανές ότι ο τραπεζικός τομέα έχει την τάση να επανέρχεται σε business as usual ε, αρκετά εύκολα, αλλά βέβαια κάτι τέτοιο δεν θα γίνει αποδεκτό ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε σε παγκόσμιο επίπεδο μετά από την κρίση. Όσον αφορά τώρα την εποπτεία και όλη τη δουλειά που πρέπει να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, είμαι πεπισμένο ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η επερχόμενη Ισπανική Προεδρία θα συνεργαστούν για να καταλήξουν σε μια στρατηγική που θα είναι αποδεκτή για όλους και θα διατηρήσει βέβαια την ε, κεκτημένη ταχύτητα της ε, προόδου που έχουμε επιτύχει. Όσον αφορά τώρα τα δημόσια οικονομικά. Είναι προφανές ότι το επίπεδο του χρέους ήταν πάρα πολύ ψηλό και μετά την κρίση ήταν προφανές ότι είμαστε σε μια κατάσταση πλέον που δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο, τα μέτρα που ελήφθησαν ήταν πολύ σημαντικά. Μιλήσαμε για 5% μείωση του ΑΕΠ, ότι θέλουμε να σταθεροποιήσουμε την ε, ζήτηση, αλλά όταν θέλουμε να έχουμε μια στρατηγική εξόδου, θέλουμε να την έχουμε γιατί αν δεν την έχουμε τα ε, μέτρα που θα λάβουμε θα είναι αποτελεσματικά μόνο βραχυπρόθεσμα. Οπότε ε, τον Οκτώβριο θέσαμε πολύ συγκεκριμένες αρχές για τη στρατηγική εξόδου ξεκινώντας ε, με την σταδιακή κατάργηση των έκτακτων μέτρων. Επίσης χρειαζόμαστε μία ε, σταθεροποίηση πάνω από το 0,5% που έχουμε αυτή τη στιγμή και επίσης χρειάζονται και κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές ε, υπέρ της ενίσχυσης της, ε, του ποσοστού ε, απασχολησιμότητας και των μακροπρόθεσμων, των μακροπρόθεσμων επενδύσεων. και η διαδικασία του Γκέτεμπουργκ αυτό το σκοπό είχε. Επίσης υπήρξε σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ε, βελτίωση του, της εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Είχαμε κάποιες συζητήσεις ε, που αφορούσαν συγκεκριμένες χώρες, εκτενείς συζητήσεις για χώρες που έχουν ε, πολύ μεγάλο έλλειμμα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή, αυτές οι χώρες αυτή τη στιγμή είναι 20. Και κατά τη γνώμη μου, Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές και από την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ειδικότερα η μακροπρόθεσμη ε, σταθερότητα που ήταν αντικείμενο μιας έκθεσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόσφατα, είναι μια μεγάλη πρόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν την, επόμενη την προβληματική κατάσταση που θα αντιμετωπίσουμε πρέπει να έχουμε βάλει μία τάξη και αυτό σημαίνει πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια ε, δημοσιονομικής φύσεως για πολλές ε, χώρες. Ε, είναι πολύ σημαντική λοιπόν η πρόκληση να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για το μέλλον. Όσον αφορά τώρα το θέμα του G20 είναι πλέον ε, το σημαντικότερο φόρουμ ε, διεθνούς οικονομικής συνεργασίας ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι το ευνοϊκό γιατί είναι σημαντικό να έχουμε μια μεγαλύτερη κλίμακα διεθνή συνεργασία λόγω της κρίσης που υπήρξε. Αλλά από την άλλη υπάρχει Δεν υπάρχει εκπροσώπηση όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην ομάδα των G20 και αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε ε, την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε όλα τα κράτη-μέλη να νιώθουν ότι μπορεί η Ευρώπη να έχει μια ισχυρή θέση γιατί θα είμαστε ισχυροί σε διεθνές προσκήνιο μόνο να έχουμε μια συντονισμένη δράση και να εισακουστεί κιόλας η άποψή μας ε, και να είναι ε, νομιμοποιημένη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγιναν λοιπόν συνεδριάσεις στο Πίτσπουργκ, στο Λονδίνο και ένα τμήμα των ε, συνεδριάσεων αφορούσε βέβαια την οικονομική ε, ενίσχυση και είναι σαφές ότι πρέπει να εφαρμόσουμε ε, στρατηγικές ε, εξόδου από τα έκτακτα μέτρα που είχαμε αναλάβει ως τώρα. Επίσης υπήρξε σημαντική πρόοδος στο πλαίσιο του G20 για την ανάπτυξη και εφαρμογή διεθνών προτύπων όσον αφορά την αποζημίωση, τη, τη λογιστική, ε, τα κεφάλαια και τη δυνατότητα ε, διάθεσης κεφαλαίων από πλευράς τραπεζών. Επίσης υπήρξε και ένα πλαίσιο ε, για ισορροπημένη ανάπτυξη που σημαίνει βέβαια ότι η διεθνή συνεργασία πλέον λαμβάνει άλλε διαστάσει. Είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία, η οποία θα συνεχίσει για κάποιο χρονικό διάστημα. Όπως γνωρίζετε ενδεχομένως ε, έγινε και πολλή δουλειά όσον αφορά τα ζητήματα κυβέρνησης από, για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, όσον αφορά την ε, εκ νέου κεφαλαιοποίηση. 125 εκατομμύρια ευρώ διέθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου δηλαδή 35% των ε, κεφαλαίων ε, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου βάσει του νέου πρόσφατου ε, διακανονισμού. Όσον αφορά τώρα τη διαχείριση των κρίσεων, υπήρξε άμεση συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν σημαντικό τμήμα της δουλειάς της Προεδρίας μας όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών. Είχαμε προβλήματα με την Ουγγαρία, την ε, Λετωνία και τη Λιθουανία που ζήτησαν ε, ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δική μας Προεδρία ασχολήθηκε κυρίως με τη Λετωνία επειδή υπάρχουν ε, και διμερείς συμφωνίες μεταξύ Λετωνίας και έξι κρατών μελών. Προσπαθήσαμε λοιπόν να ενισχύσουμε την οικονομική πολιτική της Λετωνίας αλλά επειδή ήταν πολύ υψηλό το επίπεδο της βοήθειας λόγω της οικονομικής κρίσης, ε, θα γίνει μια δεύτερη αναθεώρηση αυτή τη στιγμή και θα δούμε τι πρόοδος υπάρχει με την κατάσταση της Λετωνίας. Επίση, το θέμα του κλίματο, όπω είπα και προηγουμένω, είναι ε, ε, μία από τι βασικές μας προτεραιότητες. Η Σύνοδο Κοπενχάγη ε, άρχισε σήμερα και στο Συμβούλιο είχαμε πολλέ συζητήσει για το θέμα αυτό, γιατί υπάρχει ανάγκη συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια όταν λέω συμμετοχή εννοώ και οικονομική φύσεω. Και επίσης διαπραγματευτήκαμε μία ισχυρή ευρωπαϊκή θέση και στο G20. Αλλά βέβαια είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Είναι διαφορετικό το επίπεδο φιλοδοξία ε, που υποστηρίζουν τα διάφορα κράτη-μέλη. Οπότε υπήρχε διαφορά ανάμεσα στην κατάσταση στο Λονδίνο που ήταν κάπω απογοητευτικά τα πράγματα και κάποια, καλύτερη, κάποια πρόεδρο στο, ε, στο ε, και ενδεχομένω ακόμη καλύτερα ε, τα πράγματα στο Σαντ Άντριου παρά το γεγονό ότι δεν πετύχαμε αυτά που θέλαμε. Ελπίζουμε λοιπόν να υπάρξει πρόοδος στην Κοπενχάγη και βάσει των εκτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για παροχή σημαντικού τμήματος των πόρων που χρειάζονται αποφασίσαμε να αναλάβουμε το κομμάτι που μας αναλογεί που είναι περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουμε να επιτύχουμε την πρόοδο που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη. Πιστεύουμε ότι έχουμε την δυνατότητα ε, καλών διαπραγματεύσεων στην Κοπενχάγη, αλλά πρέπει και κάποιοι, πρέπει και οι εταίροι μας να μπορέσουν να ε, μετακινηθούν και εκείνοι κάπως από τις θέσεις τους για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό που θέλουμε. Κάτι ακόμη κοιτώντας λίγο περισσότερο το μέλλον Υπάρχει ανάγκη ανάπτυξη ε, στρατηγικών ε, για την αγορά εργασία και επειδή υπάρχουν κάποιε ιστορικέ τάσει, η στρατηγική τη Λισαβόνα θα είναι μια βασική προτεραιότητα για την επερχόμενη Ισπανική Προεδρία. Γιατί αυτό που έχουμε δει στην Ευρώπη είναι ότι κατά την περίοδο της κρίσεω αυξήθηκε η ανεργία και σιγά σιγά και αργεί πάρα πολύ να επανέλθει στα προηγούμενα τη ε, επίπεδα. Η αντιμετώπιση τη ανεργία είναι μια βασική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντική η πολιτική ανάπτυξη, αλλά η υψηλή ανεργία, η χαμηλή παραγωγικότητα ε, θα έχουν ως αποτέλεσμα ανάγκη ενισχυμένης στρατηγικής ανάπτυξης και ε, ε, καταπολέμησης της ανεργίας και γι' αυτό υπήρξαν και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του περασμένου μήνα. Όσον αφορά τα φορολογικά θέματα, στο Συμβούλιο του Νευρίου καταλήξαμε σε πολιτική συμφωνία όσον αφορά την επικαιροποίηση των ειδικών φόρων κατανάλωση για τα προϊόντα καπνού. Αυτό ήταν σημαντικό θέμα. Ήταν επιμακρών στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου. Συζητήθηκε νομίζω την πρώτη συνεδρίασή μου ως Υπουργό όταν πήγα εδώ και τρία χρόνια και ήταν στο πρόγραμμα και πριν από αυτό. Οπότε είναι μια συνεχιζόμενη ιστορία και γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλό που είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Επίσης σημειώσαμε πρόοδο όσον αφορά τον ΦΠΑ και για τις ε, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, πράσινες εκπομπές, όπου καταλήξαμε σε δυνατότητα να οι χώρες που θα χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο για να αποφύγουν απάτες όσον αφορά ΦΠΑ να χρησιμοποιήσουν αυτή τη συμφωνία μας. Θέλουμε, θέλαμε πιο φιλόδοξη ε, συμφωνία από αυτού, αλλά δεν τα καταφέραμε. Οπότε το Συμβούλιο θα πρέπει να επανέλθει όσον αφορά τα κινητά τηλέφωνα και τα ε, διάφορα, ε, διάφορες συσκευέ που έχουν ηλεκτρονικά κυκλώματα και στο ECOFIN είχα καταλήξαμε τι θα γίνει με τη φορολόγηση του ΦΠΑ για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Κάποιες χώρες όπως η Σουηδία και άλλοι έχουν την άποψη ότι είναι σημαντικό να έχουμε μια στρατηγική όσον αφορά το, την φορολόγηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών και μια σχετική οδηγία στι ταχυδρομικέ υπηρεσίε που να συμβατεί. Θα πρέπει να υπάρξει φορολογική αντιμετώπιση των ταχυδρομικών υπηρεσιών που θα ταιριάζει με την ανταγωνιστικότητα την θεμητή, το θεμητό ανταγωνισμό. Ε, καλείς ε, την Βελγική και Ισπανική ε, Προεδρία να εξετάσουν όλες τις πιθανότητες που μπορούν να εξεταστούν ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όσον αφορά αυτές τι οδηγίε. Επίσης είχα μεγάλο θέμα όσον αφορά ε, τις αποταμιεύσεις, τη δική οδηγία, όσον αφορά το πεδίο κάλυψης της οδηγίας για τις αποταμιεύσεις και να υπάρχει και πιο αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά την οδηγία αυτή για τις αποταμιεύσεις. Η πρόοδος που επετέφθη επί της οδηγίας αυτής και της οδηγίας για την διοικητική συνεργασία και την ανάκτηση ε, η συνεργασία δεν ήταν τόσο εκτεταμένη όσο ελπίζαμε και εδώ περιμένουμε η Ισπανική Προεδρία να κάνει πάρα πολλή δουλειά και να μπορέσει να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η, πρόεδρος, η Πρόεδρος. Τροφή προς και προς ερωτήσεις. Ήταν διαδικασία Catch the Eye. Όπως σας είπα, έχω έξι στον κατάλογό μου. Kay Swinburne, το πρώτο όνομα. Kay τον λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την σύνοψη των επιτευμάτων του εξαμήνου σας και νομίζω ότι υποτιμά τα μαλλιοτραβήγματα στο Συμβούλιο των τελευταίων μηνών. Είχατε τις πιο δύσκολες στιγμές και τα πιο δύσκολα καθήκοντα όσον αφορά το δημοσιονομικές ρυθμίσεις από την προκάτοχή σας. Συγχαρητήρια για τους συμβιβασμούς περάσατε το Συμβούλιο και για την πρόοδο που πετύχατε όσο αυτά τα θέματα που είχατε μπροστά σας. Όσον αφορά αυτά που αναφέρονται στα, στα πρακτικά των Συμβουλίων, για την πρόοδο που πετύχατε όσον αφορά το σώμα των εποπτών για, τη δημοσιονομική, για το δημοσιονομικό κανονισμό. Δεν προβλήθηκαν επαρκώς αυτά τα θέματα και πώς οι εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ θα λειτουργούν σε υψηλότερο επίπεδο και πώ θα υπάρξει ένα συντονισμό μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά τι χρηματοστατικέ υπηρεσίε. Τι πρόοδος έχει επιτευχθεί όσον αφορά αυτά τα θέματα του τελευταίου μήνε. Πιστεύετε ότι προχωράμε έχει αποτελματωθεί το θέμα και περιμένουμε μια γενική δομή, να δημιουργηθεί γενικότερη δομή για την εποπτεία και τον έλεγχο και να δημιουργηθεί η νέα αρχή που έχει προγραμματιστεί. Αυτά και ευχαριστώ. Υπουργό θα προτιμούσε αρκετέ ερωτήσει και μετά να απαντά. Όλε Σμιτ, επόμενο θα υποβάλει ερώτηση. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήλθατε κύριε Υπουργέ. Νομίζω <clears throat> ότι ήταν πολύ επωφελής η εργασία της ε, Σουηδικής Προεδρίας και η Επιτροπή μας πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει κάποια πρόοδος σε ό,τι αφορά τα πριμ και τα μπόνους των μάνατζερ Υπάρχουν εδώ διαφορετικά συστήματα τα οποία ισχύουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως για να έχουμε ένα ισόπεδο γήπεδο ανταγωνισμού θα ήταν καλό να υπάρχουν και παρόμοιες συνθήκες για τις ε, αποδοχές των στελεχών. Μήπως θα μπορούσε να υπάρξει και κάποια εναρμόνιση στον τομέα αυτό, να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό σύστημα για τα μπόνους και τις ε, αμοιβέ. Δεν ξέρω λοιπόν αν και εσείς ε, έχετε την ίδια άποψη με μένα. Είσαστε υπεύθυνοι επί έξι μήνες για τα θέματα του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ. Σίγουρα έχετε επιτύχει πολλά πράγματα. Στη Σουηδία θεωρεί κανείς ότι τον τελευταίο καιρό η επιρροή της Σουηδικής Προεδρίας δεν ήταν και τόσο ισχυρή. Έχετε εσείς την ίδια εντύπωση, εξακολουθείτε να είσαστε εξίσου ε, εξίσου σημαντική σε ό,τι αφορά την επιρροή που ασκείται στις άλλες χώρες ως ε, Σουηδική Προεδρία. Και ένα ακόμα ημιερώτημα ούτως πίν που θέλω να σας απευθύνω. Πιστεύετε ότι τώρα θα μπορεί η Σουηδία κάποια στιγμή να μπει πια επιτέλους στη ζώνη του ευρώ ή όχι. Ή όχι. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, λέει ο κύριος Λάγκεν. Ήταν <clears throat> εκτελής ο απολογισμός που κάνατε. Ήταν σίγουρα για μια μεγάλη χώρα όπως η Γερμανία ένας πολύ θετικός απολογισμός. Παρ' όλα αυτά θέσατε πολλά ερωτήματα Είπατε ότι σε μεγάλο βαθμό έχει ξεπεραστεί η κρίση. Επιτρέψτε μου να τρέφω σοβαρέ επιφυλάξει για κάτι τέτοιο, για το αν η κρίση αυτή έχει πράγματι υπερπηδηθεί. Για να γίνει κάτι τέτοιο για μένα είναι απαραίτητο σε ό,τι αφορά τον, ε, ε, την εποπτεία των χρηματαγορών να βελτιωθεί σημαντικά η απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα ισόπεδο γήπεδο για τον ανταγωνισμό και ίσες συνθήκες για όλους. Το δεύτερο σημείο το οποίο θέλω να σας θέσω υπομορφή ερωτήματο ερωτήματος είναι το θέμα της στρατηγικής εξόδου. Μπορώ να κοιτάξω την Ελλάδα, τη Γερμανία ή την Γαλλία και έχω πολλές αμφιβολίες ότι υπάρχει κάποια στρατηγική εξόδου από τα πολύ υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα των χωρών αυτών. Θα ήμουν ευγνώμα αν μπορούσατε να μου εξηγήσετε με ποιο τρόπο θα μπορέσει να είναι επιτυχής μια τέτοια στρατηγική εξόδου. Τρίτος τομέας σε ποιο βαθμό επιτύχατε φέτος στην, ε, στα θέματα των χρηματαγορών να καταλήξετε σε συμφωνία με τις Αμερικανικές αρχές. Ανεφέρθη ο κύριος Σμιτ στο σύστημα των πόνους για τα στελέχη και βλέπω ότι στις ΗΠΑ υπάρχει μια πάρα πολύ έντονη συζήτηση γιατί η Goldman Sachs θα δώσει 21 δισεκατομμύρια δολάρια bonus. Είναι το μεγαλύτερα, τα μεγαλύτερα bonus στην ιστορία των επιχειρήσεων αυτών. Πώς μπορεί να γίνεται σε μια εποχή κρίσεων να δίνει τόσο υψηλά bonus μια επενδυτική τράπεζα. Είσαστε έτοιμοι να αναλάβετε κάτι για να αντιμετωπίσετε τα θέματα αυτά και το τελευταίο ερώτημά μου το έθεσε ήδη ο κύριος Σμιτ. Θα χαιρόμασταν πάρα πολύ αν επιτέλους κάνει το βήμα η Σουηδία και μπει στη ζώνη του ευρώ. Είσαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Τι άλλο χρειάζεται για να σας οδηγήσει στη ζώνη του ευρώ. Γιατί αντίθετα από τη Μεγάλη Βρετανία και τη Δανία δεν έχετε κάποια ρήτρα opt-out αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις σκέψεις, τα σχόλια. Όσον αφορά το ερώτημα της Σουηδίας για το σώμα των εποπτών, των εποπτικών αρχών, Δώσαμε ύψιστη προτεραιότητα στην μικρο και μακροεποπτεία στα πλαίσια της δομής που δημιουργήθηκε επί Προεδρίας μας. Βασικά χαρακτηριστικά αυτά είπατε βέβαια ότι έπρεπε να ήμασταν πλέον φιλόδοξοι. Νομίζω ότι πετύχαμε κάνα δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε τη βάση για μια δομή και από πλευράς μακροεποπτείας και μικροεποπτείας. Δεύτερον, καταφέραμε να κάνουμε σωστό ξεκαθάρισμα των στοιχείων. Όταν ξεκινήσαμε στην Προεδρία μας, το πρώτο θέμα θέσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αν θα μας υπέβαλαν αρχή Σεπτεμβρίου νομοθετική πρόταση. Το έκαναν οι απ' σχολιαστές, έλεγαν δεν είναι δυνατόν, δεν μπορούν να κάνουν σε λίγους μήνες προπαρασκευαστική εργασία. Διότι πήραμε απόφαση στο Συμβούλιο μόνο αρχές του καλοκαιριού. Οι περισσότεροι μας είπαν όταν στο Γκέτεμπορκ είπαμε ότι πρώτα θα εξετάσουμε τη μακροεποπτεία και μετά τη μικροεποπτεία επί Σουηδικής Και τα ΜΜΕ έλεγαν ότι αυτό ήταν υπερβολικά φιλόδοξο, δεν ήταν ρεαλιστικό να πετύχουμε συνένεση επί των δύο θεμάτων Οκτώβριο και Δεκέμβριο. Τα καταφέραμε όμως. Και κρατήσαμε ενωμένη την Ευρώπη παράλληλα. Όλοι έχουμε ευθύνη να έχουμε μια συνεκτική Ευρώπη, όπου όλα τα κράτη-μέλη να αισθάνονται ότι το σύστημα λειτουργεί για όλους. Σέβομαι όσους λένε ότι βεβαίως έχω βεβαίω ιδιαίτερο συμφέρον ή όπως τα βλέπει η χώρα μου θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερη λύση. Ναι, αληθεύει ίσω, διότι μιλάμε για συμβιβασμό εδώ. Θέλαμε να έχουμε αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που να δέχονται όλοι και να είναι και αρκετά αισιόδοξο ο στόχο. Έτσι δουλεύει η πολιτική. Πάντα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα και να προσπαθούμε να συγκεράσουμε τα συμφέροντα και να βρούμε ισορροπίε. Θα υπάρξει καλό αποτέλεσμα από τις προσπάθειες Κοινοβουλίου, Ισπανικής Προεδρίας και Συμβουλίου για να επεξεργαστούμε το συμβιβασμό. Συμβιβασμός είναι. Δεν μπορούμε να έχουμε μια λύση που είναι τέλεια για μα, αλλά δεν είναι καλή για τα άλλα κράτη-μέλη. Πρέπει να βρούμε κάτι που είναι καλό για όλη την Ευρώπη. Και ποιο είναι το μάθημα που αποκομίζω από την κρίση. Χρειάζεται μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συνεργασία, ισχυρότερη ευρωπαϊκή θεσμή, περισσότερε κοινέ λύσει. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι ξεκάθαρο ο δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Τι ρυθμό θα ακολουθήσουμε όμω. Όλοι ε, εκπροσωπούμε μεταρρυθμιστικές παραδόσεις. Πρέπει να μεταρρυθμίζουμε με έναν τρόπο τέτοιο που να εξακολουθεί να συνεργάζεται αγαστά η Ευρωπή. Ο κ. Σμιτ αναφέρθηκε στον κανονισμό τη διαθέτηση των μπόνους. Το ανέφερε ο κ. Λάγκεν. Ναι, παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν αρκετέ διαφορέ, σημαντικέ διαφορέ μεταξύ χωρών. Σουηδία, Γαλλία, Ενωμένο Βασίλειο ήδη αρχίζουν να εφαρμόζουν τι αποφάσει που ελήφθησαν στο Pittsburgh και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες που δεν ξεκίνησαν καν τη διαδικασία. Πολύ προβληματικό αυτό. Επίσης, έγινε δήλωση όλων των Ευρωπαίων ηγετών που υποστηρίζουν διαδικασία συντονισμού ότι είναι βασική αρχή που θα πρέπει να χρησιμοποιούμε, ότι θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση, θα παρακολουθεί το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αυτό το ζήτημα και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τεθεί στο Συμβούλιο. Εάν στον τραπεζικό τομέα κινηθούμε σαν να μην τρέχει τίποτα, κάτι που υπονόησε το ερώτημα του κ. Λάγκενς, θα ακολουθήσει και περισσότερη ρύθμιση. Αυτό θα ήταν απαράδεκτο και σε επίπεδο Ευρώπης και σε επίπεδο G20. Φαντάζομαι, προβλέπω, ότι ε, θα, υπάρξουν απαράδεκτες πρακτικές για μπόνους στην Άνοιξη, θα χρειαστεί και άλλος γύρος διεθνών πολιτικών συζητήσεων για τα μπόνους και αυτό σημαίνει ότι στο, μέλλον θα πρέπει να, στο μέλλον θα πρέπει να γίνει πιο αυστηρός ο σχετικός κανονισμός για τα μπόνους. Τώρα το ερώτημα του κυρίου Σμιτ για το ECOFIN και το Eurogroup και τον συντονισμό τους. Κοιτάξτε, πολύ καλή συνεργασία με τις χώρες της Ευρωζώνης και το Eurogroup α το πούμε ξεκάθαρα, συζητήσει για το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη έγιναν και στο ΕΚΟΦΗΝ και στο Eurogroup. Αρκετέ φορέ η συζήτηση εστράφη, μάλλον συζητήθηκαν περισσότερο τα θέματα στο ΕΚΟΦΗΝ από ότι στο Eurogroup. Σημαντικό θεσμό και το Eurogroup θα πρέπει να διεξαγάγει και εκεί συζήτηση διεξοδική για το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη αλλά εκεί μέχρι τώρα το ECOFIN διαδραμάτισε σημαντικότερο ρόλο όσον αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη από το Eurogroup. Τώρα, αν μπει στο ευρώ, η Σουηδία θα είναι πρόοδο, ναι. Αυτό πιστεύω. Να μπούμε το ταχύτερο να απάντηση, ναι. Σημαίνει αυτό ότι μπορούμε να έχουμε και υποστήριξη σε δημοψήφισμα στη Σουηδία για να μπούμε στην Ευρωζώνη. Υπάρχει σαφής δήλωση όλων των ηγετών των κομμάτων που υποστηρίζουν το ευρώ ότι θέλουν δημοψήφισμα. Και στο δημοψήφισμα που διεξήχθη ήταν φανερό ότι χρειάζεται χρόνος μέχρι να ξανατεθεί το θέμα μέσω δημοψηφίσματος. Θα μπούμε στο ευρώ όσο όποτε μπορούμε, αλλά το θα μπορούμε να μπούμε, το θα μπορούμε σημαίνει ότι θα πρέπει να μπορεί να περάσει και το δημοψήφισμα. Θα είναι καλό και για τη Σουηδία και για τις άλλες χώρες. Οι χώρε είναι σε καλύτερη θέση με το ευρώ παρά χωρί το ευρώ, πιστεύω. Ο κ. Λάγκεν ρώτησε κατά πόσο Έχουμε βγει από την κρίση. Προφανώ αυτό εξαρτάται πώ το βλέπει, από την οπτική γωνία από την οποία βλέπει. Ξαναδουλεύουν οι τραπεζικέ αγορέ, οι πιστώσει αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δεν τόσο άσχημα τα πράγματα τώρα όσο ήταν πριν από ένα εξάμεινο όμω. Πρέπει να θυμηθούμε ότι το Φεβρουάριο-Μάρτιο μόλι βλέπαμε μελέτε που συνέκριναν την κατάσταση αυτή με τη δεκαετία του 30 που είχαμε αρκετά χρόνια τότε αρνητική ανάπτυξη και ανεργία είχε χτυπήσει το 15 20% στην Ευρώπη ο κίνδυνος τέτοιων εξελίξεων τώρα πλέον εξέλιπε. Κάναμε αρκετά για να βγούμε από την κρίση. Με καλύτερη οικονομική, ε, χρηματοπιστωτική δομή. Ναι. Η βελτίωση είναι αρκετή. Α, αυτό πρέπει να το εξεργαστούμε, να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι καλό ήταν ότι πήραμε αποφάσεις γρήγορα, διότι διαφορετικά οι ψηφοφόροι και η εμπιστοσύνη του κόσμου θα έχει υπονομεθεί στην Ευρώπη, θα λέγανε ότι οι πολιτικοί ηγέτε ε, δεν πήραν τι σωστέ αποφάσει και δεν έμαθαν τα μαθήματά του από την κρίση. Όσον αφορά την στρατηγική εξόδου για δημοσιονομική πολιτική, εγώ εκπροσωπώ μια χώρα που θέλει σε δύο-τρία χρόνια να μπει πάλι σε πλεόνασμα. Εγώ δεν θα, ε, δεν θα πρότεινα 3% έλλειμμα Αυτό το κριτήριο ελλείμματο 3% του συμφώνου σταθερότητα και ανάπτυξη είναι πολύ περιορισμένο. Εγώ θα έλεγα πριν μπούμε στην επόμενη κρίση να, βγουν, να μπουν στην ανάκαμψη χώρε. Το σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη τι λέει 3%. Στι αρχέ τη Ουδική Προεδρία έγιναν πολλέ συζητήσει κατά πόσο μπορούμε να καθορίσουμε κάποιε αρχέ. Αν μπορεί να υπάρχει δίκαιη αντιμετώπιση των χωρών. Και αρχέ που καθορίστηκαν στο Γκέτεμποργκ που ήταν βάση για αποφάσεις και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και με τι διαδικασίε υπερβολικού ελλείμματο, οι αποφάσει που ελήφθησαν ήταν σημαντικό βήμα πρόοδο. Αλλά χρειάζεται να είμαστε πιο φιλόδοξοι όσον αφορά τη δημοσιονομική πολιτική στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Κάρις, Κιούρις και Λουτβίντσεν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε για το δημοψήφισμα που αφορά το ευρώ. Εγώ χαίρομαι που θέλετε να μπείτε το ταχύτερο να στη ζώνη του ευρώ η Σουηδία. Είπατε ότι στη χώρα σας ζητούν τα πολιτικά κόμματα να υπάρχει ένα δημοψήφισμα. Αλλά πότε, αν όχι τώρα, δεν είναι κατάλληλη στιγμή να κερδίσετε τον πληθυσμό σε ένα δημοψήφισμα υπέρ του ευρώ, τη στιγμή που το ευρώ ήταν η καλύτερη ασπίδα για τη χρηματοοικονομική και οικονομική κρίση. Επίσης, αναφερθήκατε στην εποπτεία των ε, χρηματαγορών. Εδώ το ερώτημα είναι πάλι ένα θέμα προοπτικής. Το Συμβούλιο αποφάσισε λιγότερο από αυτά τα οποία πρότεινε η Κομισιόν, που είναι λιγότερα από αυτά που θέλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, λιγότερα από αυτά που θέλει η Επιτροπή Δελαροζία, λιγότερα από αυτά που ήθελε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν λέτε για συμβιβασμό, είναι συμβιβασμός μεταξύ των κρατών ε, μελών, αλλά δεν υπάρχει συμβασμός μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς λέμε ναι να υπάρχει και μακροοικονομική και μικροοικονομική εποπτεία, αλλά χρειαζόμαστε πραγματικά να υπάρχουν αρμοδιότητες για την εποπτεία αυτή και δυνατότητες κυρώσεων. Μόνο όταν τα δεχτείτε αυτά μπορούμε να κατα... μπορείτε να καταλήξετε σε μια συμβιβαστική λύση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, το θέμα των hedge funds, hedge funds το Συμβούλιο και πάλι δέχτηκε πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία είχε ζητήσει η Κομισιόν, παρά το γεγονός ότι εμείς έχουμε πια το δικαίωμα της συναπόφασης. Και θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια λύση χωρίς την συναπόφαση του Κοινοβουλίου, ιδίω αν υπολείπεται πόρο της πρότασης της Κομισιόν. Θα ήθελα λοιπόν να σκεφτείτε και να αντλήσετε και συμπεράσματα από τη νέα αυτή κατάσταση που θα προκύψει με την δυνατότητα συναπόφαση από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Και εγώ θέλω να σας συγχαρώ για τον τρόπο με τον οποίο συνοψίσατε τις επιτυχίες και τις προσπάθειες της ε, Σουηδικής Προεδρίας. Θέλω να σταθώ στο θέμα των φορολογικών, των λεγόμενων φορολογικών παραδείσων. Στη διάσκεψη κορφής των G20 είχαν αναφερθεί και είχαν γίνει υποσχέσεις για έντονους περιορισμούς των φορολογικών παραδείσων και όλες οι χώρες είχαν δεχθεί να δίνουν στοιχεία για αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους. Τώρα, θεωρείτε ότι επαρκούν τα τωρινά πρότυπα του ΟΣΑ για να αντιμετωπιστεί το θέμα των ε, φορολογικών παραδείσων. Υπήρξε μια συμφωνία και 12 κρατών για την ανταλλαγή παρα... πληροφοριών σε σχέση με τους φορολογικούς παραδείς... παραδείσους. Μπορεί να αυτό όμως να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και ποια μέτρα θεωρείτε ότι πρέπει να ληφθούν περαιτέρω. Επίσης υπάρχει συζήτηση μέσα στο Συμβούλιο ότι σε περιπτώσεις προμηθειών δημοσίων θα μπορούν να συμμετέχουν μονάχα οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμπλέκονται με φορολογικούς παραδείσους. Υπάρχουν και εδώ νέες σκέψεις από την πλευρά του Συμβουλίου ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ ιδιαίτερη χαρά μας να σας έχουμε μαζί μας. Είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση με τον κύριο Τρισέ, ο οποίος μας είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η κατάρτιση για τη μείωση της ε, ανεργίας. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη μείωση του αντικτύπου της κρίσης, ειδικότερα σε μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση, όπως η ευρωπαϊκή οικονομία. Στη Σουηδία, έχουμε 40% λιγότερη επαγγελματική κατάρτιση από ότι το 2006. Και πρέπει η κατάρτιση να απευθύνεται περισσότερο σε εκείνους που τη χρειάζονται για να επανέλθουν στην αγορά εργασίας. Το Συμβούλιο προτείνει περικοπές στα μέτρα κατάρτισης. Εσείς συμφωνείτε. Ποια είναι η άποψη της Προεδρίας για τη χρηματοδότηση από πλευράς κοινότητας των μέτρων αυτών κατάρτισης. Και όσον αφορά το ευρώ, ναι, και, εμείς, και εγώ συμφωνώ, οπότε σε αυτό συμφωνούμε. Υπουργό, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά το θέμα του, που έθεσε ο κύριος Κάρας για το δημοψήφισμα στη Σουηδία, υπάρχει κάτι που πρέπει να τονιστεί. Η Σουηδία δεν είναι εκτός ευρωζώνης ε, για να έχει λιγότερο υπεύθυνη οικονομική πολιτική. Έχουμε ένα στόχο για τον πληθωρισμό και μάλιστα θα έλεγα ότι είχαμε και χαμηλότερο πληθωρισμό, μέσο πληθωρισμό, από πολλές χώρες της Ευρωζώνης. Όσον αφορά τώρα τους δημοσιονομικούς μας στόχους, είναι πολύ αποτελεσματικοί και κρίνεται αυτό και από τα αποτελέσματά τους σε σχέση με την Εστονία, τη Βουλγαρία, ε, που είναι, έχουν πολύ υψηλό δημοσιονομικό χρέος, έλλειμμα, συγγνώμη. Όσον αφορά το συγκλητικό πλεονέκτημα του να μην συμμετέχει κανείς στην Ευρωζώνη, εγώ διαφωνώ με αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα αν θέλουμε να επιτύχουμε οικονομική σταθερότητα εκτός Ευρωζώνης. Ε, εντάξει, η Σουηδία μπορεί να έχει λιγότερε συνέπειε από την κρίση, αλλά ήταν σοβαρά τα προβλήματα και με την ανάπτυξη και με την ανεργία στη Σουηδία λόγω της κρίσεως. Επομένως, ελπίζουμε να έχουμε σύντομα την υποστήριξη του σουηδικού λαού. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τους πείσουμε και τότε θα προσπαθήσουμε να μπούμε στην Ευρωζώνη. Όσον αφορά το θέμα της συναπόφασης με το Κοινοβούλιο, θα ήθελα να τονίσω Ε, είναι, ήταν για μας λίγο προβληματικό το γεγονός ότι δεν είχαμε όλα τα στοιχεία ακόμη στη διάθεσή μας ε, λόγω της κατάστασης με τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, και εμείς υποστηρίξαμε τις προσπάθειες της Σουηδικής Προεδρίας να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ένας συμβιβασμός, κάποιες παναχωρήσεις και από, πλευρά, και από πλευράς του Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι σε μεγάλες αποφάσεις ε, πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ευρία συνένεση, να λάβουμε υπόψη ολόκληρο το πολιτικό σφάσμα όσο το δυνατόν ε, μπορούμε. Νομίζω ότι μόνο έτσι θα έχουμε μια ε, πραγματική Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχυρότερη. Θα είναι περίπλοκες οι συζητήσεις με το Κοινοβούλιο γιατί είναι ένα περίπλοκο ζήτημα αυτό από πολλές απόψεις. Όσον αφορά τα hedge funds, ε, θυμόμαστε όλοι τι έγινε το 1998 όταν τα μακροπρόθεσμα κεφάλαια ε, απέτυχαν και θυμάστε τότε τι έγινε και με τη ε, ρωσική οικονομική κρίση. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να υπάρχει κάποιο είδους εποπτεία και γι' αυτό συμφωνώ ότι μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο και πρέπει να υπάρξει και συνένεση προς αυτή την κατεύθυνση. Με ρωτήσατε για τους φορολογικούς παραδείσους. οι αποφάσεις που λάβαμε στο Λονδίνο έχουν εφαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό. Δεν υπάρχουν ε, σε ε, γκρίζες λίστες πλέον ε, χώρες. Έχει υπάρξει πολύ σημαντική πρόοδος σε σχέση με τους φορολογικούς παραδείσους. Τώρα, εμείς ως Σουηδία ενδιαφερόμασταν πάρα πολύ γιατί θεωρούμε ότι χάνουμε πάρα, πάρα πολύ φορολογικό εισόδημα όπως και άλλες χώρες και γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να σημειωθεί πρόοδος. Δεν πρέπει βέβαια να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι έχει ήδη υπάρξει κάποια πρόοδος. Και η Ισπανική Προεδρία πρέπει να ασχοληθεί και με το θέμα της οδηγίας για την αποταμίευση. Να υπάρχει αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, και να έχουμε και σοβαρές συζητήσεις με πολλούς γειτονές μας για το θέμα αυτό. Τώρα όσον αφορά το θέμα που έθεσε ο Σουηδός συνάδελφος για την κατάρτιση, εγώ δεν βλέπω να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη δική μου θέση, τη θέση της Σουηδικής Προεδρίας και της άποψης του κυρίου Τρισέ. Πιστεύουμε ότι η κατάρτιση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που προσπαθήσαμε να προωθήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια ε, της Προεδρίας. Στο Γκέτερμπουργκ ε, ένας από τους βασικούς εμπειρογνώμονες ε, τη της ε, αγοράς εργασίες, εργασίας ε, ε, μας υπέβαλε την άποψή του και ο κύριος Αλμούνια έχει σημαντική εμπειρία στον τομέα αυτό λόγω της εμπειρίας του στην Ισπανία αλλά είναι γεγονός ότι Εκτός από την κατάρτιση μπορεί να υπάρχει και η, δυνατό, η διευκόλυνση των ατόμων να βρουν ε, κάποια εργασία, κάποια μέτρα ενεργά κατά τη διάρκεια της ε, περίοδου της ανεργίας. Νομίζω λοιπόν ότι η κατάρτιση είναι ένα σημαντικό ε, τμήμα της αντιμετώπισης της κρίσης και μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, αν θέλουμε να αυξήσουμε την κοινωνική συνοχή, νομίζω ότι ε, η κατάρτιση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τέσσερις ακόμη έχουν μείνει στον κατάλογο των ομιλητών και θα τους ακούσουμε όλους. Σβέν. Well, I, I have... Έχω δύο διαφορετικά ερωτήματα, τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους. Καταρχήν, φορολογική παράδειση και οδηγία για την αποταμίευση. Μπορείτε να μας εξηγήσετε ποια ήταν τα επίμαχα σημεία και ποιες χώρες τι πήρανε ποια θέση και γιατί αυτό μας οδήγησε σε μια κατάσταση αδυναμίας συμφωνίας κατά τη διάρκεια της πρόεδρης. Θέλω να έχω κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες δυνατόν. Δεύτερον, για το θέμα του χρέους, του δημοσίου χρέους ορισμένων κρατών μελών. Βλέπουμε υψηλά και ανησυχητικά επίπεδα δημόσιου χρέους. Λέτε όμως συγχρόνως, και συμφωνώ μαζί σας, ότι χρειαζόμαστε περισσότερη δημοσιονομική συνεργασία στην Ευρώπη. Υπήρξαν συζητήσεις, υπήρξε πρόοδος για το πώς θα διαρθρωθούν όλα αυτά πώς θα υπάρξει μεγαλύτερη ολοκλήρωση στην ευρωπαϊκή οικονομία και πόσο μακριά έχουμε φτάσει με συνεργασία για να μπορέσουμε να έχουμε κοινό επίπεδο φορολογίας ώστε και οι χώρες να έχουν επίσης χαμηλότερα επιτόκια τα οποία πρέπει να πληρώνουν για την εξυπηρέτηση του δημοσίου τους χρέους. Τι έχει συζητηθεί λοιπόν σχετικά για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν το χρέος τους και να το μειώσουν καιρό η Κάθριν Στάιλερ. Ναι, κάτι λάθος έχω κάνει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και τον κύριο Υπουργό για την παρουσίασή του επίσης. Τρία σημεία. Καταρχήν ο φόρος στις ε, χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Είχαμε διοργανώσει μια ενδιαφέρουσα ακρόαση στην Επιτροπή μας και ποια είναι η αποψή σας για το θέμα αυτό φορολογίας για τις ε, χρηματοοικονομικές συναλλαγές και πώς θα μπορούσατε εσείς να ορίσετε ένα τέτοιο φόρο. Για το θέμα των πόνους επίσης, κάτι το οποίο αναφέρθηκε σε μια συνάντηση που είχαμε συνδικαλιστές την προηγούμενη ε, Παρασκευή στον, στην εκλογική μου περιφέρεια. Συνδικαλιστές από τον τραπεζικό τομέα. Είπαν ότι υπάρχουν άτομα τα οποία δεν είναι σε διευθυντικές θέσεις, που εργάζονται πολύ σκληρά, που είναι στις τράπεζες 20 χρόνια και παραπάνω και δεν λαμβάνει κανείς υπόψη <clears throat> την οικονομική κρίση όταν ε, αξιολογούν την απόδοσή τους, θεωρούνται ότι δεν αποδίδουν και επομένως τους απολύουν στη συνέχεια. Μια τράπεζα έχει κάπου 10% του προσωπικού της σε κατάσταση που ζητούν αυτή τη στιγμή να δικαιολογηθεί η απόλυσή τους. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα λοιπόν, όχι μόνο στι τράπεζε, αλλά και άλλοι εργαζόμενοι που είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Οι άνθρωποι λοιπόν που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση αναγκάζονται να εργάζονται με μερική εργασία. Είναι γυναίκε που γυρίζουν από μία άδεια μητρότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι, ακόμα και μέσα στον τραπεζικό τομέα. Μήπω συμφωνείτε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει μια νέα μορφή εταιρικής ευθύνης, ένα νέο υπόδειγμα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες για να έχουμε μια καλύτερη ισορροπία. Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι θα πρέπει τα μπόνουσες να καταργηθούν και όχι κάτι το οποίο θα είναι αντικείμενο συζήτηση στην Επιτροπή μας. Και όταν μιλάτε για εκατομμύρια σε μπόνους, ενώ άλλα άτομα μετά από 20 χρόνια εργασίας τους δίνουν αποζημίωση τριών μηνών. Πώς μπορούμε να τα συμβιβάσουμε όλα αυτά τα θέματα. Και επίσης η λογιστική ε, δίκαιου τιμήματος για τις μετοχέ. Αναρωτιέμαι αν έχετε κάποιες προτάσεις για το θέμα αυτό για να εφαρμοστούν λογιστικά πρότυπα αυτού του είδους. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας και τον χρόνο σας. Κύριος Σάιμον, το ερώτημά μου και εμένα αφορά πάλι το θέμα της ευρωπαϊκής ε, εποπτείας και επίσης το κατά πόσο αυτή μπορεί να συμβιβαστεί με τις εθνικές αρχές. Εγώ νομίζω, βλέπω εδώ ότι έχετε μια τετραπλή διαδικασία. Έχουμε τις ε, εθνικές ε, αρχές, έχουμε τις ευρωπαϊκές αρχές και στη συνέχεια το ερώτημα είναι ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία για να αντιληφθούν μέτρα, αλλά το εθνικό κράτος έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει και να εγείρει μια ένσταση. Και μετά υπάρχει ένας χρονικός, ένα χρονικό διάστημα άλλων δέκα ημερών για να εξεταστεί αυτό και τότε μονάχα έχει ένα κράτος το δικαίωμα να προσφύγει στο, Ευρωπαϊκό, στο Συμβούλιο των Υπουργών. Βλέπετε λοιπόν τι γίνεται όταν περνάει ο χρόνος μέρα με τη μέρα, <clears throat> όπως έγινε στην περίπτωση της κρίσης και δεν υπάρχει δυνατότητα μια ταχεία αντίδρασης. Αυτό λοιπόν δεν οδηγεί, αυτό το σύστημα που προβλέπεται δεν οδηγεί σε πιο μακρού χρόνου, και αυτό δεν μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε σωστά μια κατάσταση κρίσης. Um, um, Έχω άλλους δύο. Vicky Ford και Astrid Λοιπόν, πρώτα τις τρεις να απαντηθούν οι τρεις ερωτήσεις και μετά ακολουθούν οι άλλοι δύο. Ευχαριστώ, λέει ο Υπουργό για τα ενδιαφέροντα ερωτήματα, ξεκινώντας με το πρώτο ερώτημα για τους φορολογικούς παραδείσους και το έργο της οδηγίας περί αποταμιεύσεων πρέπει να πω ότι οι λύσει και συμβιβασμός είναι εφικτά. Είμαι Σουηδός, άρα εγώ πιστεύω βέβαια πως καταλαβαίνετε συμβιβασμούς θα μπορούσαμε, πιστεύω, να καταλήξουμε σε συμβιβασμό όσον αφορά την οδηγία περί αποταμιεύσεων αν είχαμε άλλε μία ή δύο συνεδριάσεις διότι υπήρχαν πολλά τεχνικά περίπλοκα ζητήματα παρέμειναν εκκρεμή και επειδή ήταν μακροσκελέστατη διαδικασία για τα υποπτικά ζητήματα δεν κατέστη δυνατόν να ξεκινήσουν τόσο περίπλοκες διαπραγματεύσεις με πετυχημένα αποτελέσματα στην τελευταία συνεδρίαση του ΕΚΟΦΗΝ θα πρέπει να είναι έτοιμες κάποιες χώρες να κινηθούν λίγο πιο πέρα. Βεβαίως μιλάμε για ισορροπία. Θέλουμε να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής οδηγίας για τις αποταμιεύσεις. Ε, υπάρχουν διάφορα σημεία που είναι εκτός πεδίου εφαρμογής της οδηγίας και πρέπει να καλύπτονται. Θα πρέπει να προχωρήσουμε βάσει τη συμφωνία του Φιέρα του 2002 ε, όσον αφορά την εφαρμογή του συστήματος αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών Χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία το ζήτημα. Δεν θα πρέπει να υποτιμά κανεί το βαθμό των προβλημάτων και αμφιλεγωμένων ζητημάτων. Εγώ πιστεύω ότι μπορούν να επιληθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα οι διαφόρες. Ε, θέλουν πολλοί τα κράτη-μέλη να σημειωθεί η πρόοδο. υπαρχουν Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που έχουν επιφυλάξει επιφυλάξεις, πολύ γνωστά κράτη-μέλη, επί αρκετών οδηγιών που αφορούν τον τομέα αυτό αλλά τεχνικές συζητήσεις οι χώρες αυτές ήδη ανέφεραν ότι είναι έτοιμες να συνεργαστούν προς εξέβρεση λύσεως. Όσον αφορά το επίπεδο χρεώσεως δεν εξαρτάται από την οπτική γωνία ε, που ακολουθεί σε αυτά τα οικονομικά θέματα. Ε, το χρέος και το έλλειμμα είναι θέματα που πρέπει να ελπιδηθούν. Όταν μιλάμε για θέσεις ε, και οικονομικές κρίσεις πρέπει να έχουμε μια αφετηρία Πριν μπούμε στη νέα ύφεση ε, με ισχυρότερες χρηματοδοτήσεις από πλευράς του δημόσιου τομέα, μιλώντας από ειδική πλευρά. Όταν έχεις μεγάλο έλλειμμα, χρειάζονται σοβαρές αποφάσεις, όχι μόνο για τους φόρους, αλλά για τις δαπάνες επίσης Υπάρχουν φόροι και δαπάνες που επηρεάζουν επικοινωτρόπο την κοινωνική συνοχή, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Έχουμε τον φόρο επί του άνθρακος, καλός για το περιβάλλον. Έχουμε φόρους για τα καύσιμα, για τον καπνό, για το ενόπνευμα που δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς στην Ευρώπη ε, και θα μπορούσαν να αυξήσουν τους δημόσιους πόρους χωρίς να πλήξουν την ανάπτυξη. Έχουμε δαπάνες σημαντικότητες για την ανάπτυξη, επενδύσεις για υποδομές κλπ αλλά υπάρχουν και δαπάνες που σε μεγάλο βαθμό είναι αποτελέσματα μη δυνατότητας να κρατήσουμε κόσμο στην αγορά εργασίας. Όσον αφορά τις δαπάνες χρειαζόμαστε πάρα πολύ υπεύθυνε προσπάθειες αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την χρέος, το χρέος. Η Κάθριν Στήλερ έθεσε το ερώτημα για το φόρο οικονομικών συναλλαγών, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Εγώ υπέβαλα πρόταση και λήφθηκε απόφαση στη Σουηδία, πρόταση να ε, ζητείται ένα τέλος από πλευράς τραπεζών ανάλογα με το μέγεθος του ισοζυγίου τους. Ε, είχαμε έναν φόρο συναλλαγών, δεν λειτουργήσε γιατί περισσότερε συναλλαγές είναι πάρα πολύ ρευστές και σε μεγάλο βαθμό εκκινούνται εκτός της ε, δικής μας δικαιοδοσίας. Ένας φόρος όσον αφορά το ισοζύγιο αυτό είναι κάτι πολύ πιο περίπλοκο προ αποφυγή, διότι χρειάζεται ισοζύγιο και έχουμε πάρα πολλέ ισχυρέ διευθετήσει και νόμου όσον αφορά το υποπτικό και ρυθμιστικό έργο στον τομέα των τραπεζών, το ισοζύγιο των τραπεζών και για να πούμε ειλικρινά, αν έχουμε πρόβλημα χρηματοστικής αστάθεια ή δημιουργίας ε, νέου ομφόλιγα, θα πρέπει να το δούμε τι γίνεται όσον αφορά την επέκταση κάλυψης του ισοζυγίου των τραπεζών. Εμεί φορολογούσαμε ένα τέλο, τέλο, δεν είναι φόρο. εισπράταμε ένα τέλο, λοιπόν, για να διευκολύνουμε ένα ταμείο, να τροφοδοτούμε ένα ταμείο σταθεροποίησεως που στο μέλλον θα αντιμετώπιζε τα προβλήματα του τραπεζικού τομέα. Γιατί θα ήταν σωστό να πληρώνει για την ασφάλισή του ο ίδιο ο τραπεζικό τομέα. Και υπάρχουν αρνητικέ συνέπειε για ένα μεγάλο αρνητικό. Ε, αρνητικές συνέπειες για μεγάλο τραπεζικό τομέα πρέπει να εξεταστεί. Καταλαβαίνω εκείνου που συναντήσε η Κάθριν Στήλερ, άνθρωποι του τραπεζικού τομέα που εργάστηκαν ε, με πίστη προς την τράπεζά τους σε μεγάλο χρονικό διάστημα και χωρίς να φταίνε αυτοί αντιμετωπίζουν την ε, πολύ σοβαρή κρίση. Όμως ταυτόχρονα βλέπουμε και πάρα πολύ μεγάλα μπόνους που δίνουν σε ε, ανώτερα στελέχη αυτών των τραπεζών. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το τραπεζικό θέμα και το θέμα των μπόνους σωστά. Λοιπόν, αν δεν θέλουμε να παίρνουν, αναλαμβάνουν κινδύνους ε, ο κόσμος, δεν θα γίνουν οι σωστές κινήσεις και δεν θα πρέπει όμως να κινδυνεύουν να αντιμετωπίσετε κίνδυνος μέσω τεραστίων ποσών που διατίθενται για να βοηθήσουμε τις τράπεζες. Πρέπει να υπάρχει σωστή, σωστό συνέστημα ευθύνης και σωστής αντιμετώπισης. Και κάποια λόγια να πω τώρα όσον αφορά τα προβλήματα που έφυξε ο κ. Σίμων. Αν θέλουμε πιο φιλόδοξες προπτικές, λιγότερο φιλόδοξες προπτικές όσον αφορά το χρηματοστικό τομέα και δημοσιονομική πολιτική. Δεν θα πρέπει να υποτιμάμε τι αντιμετωπίζουμε εδώ πέρα. Είναι ε, 2-3% του ΑΕΠ κόστησε στη Σκανδιναβία αυτή η τραπεζική ε, κρίση ήταν πιο φθηνή. Ε, λιγότερο από 60% του ΑΕΠ ήταν στην Ονησία. Ήταν πιο ακριβό το κόστος. Και οι υπόλοιποι πλήρωσαν ένα τίμημα ανάμεσα στα δύο άκρα. Τεράστιο ο κίνδυνο αντιμετωπίζει η δημοσιονομική πολιτική. Ιστορικά είδαμε διαφορετική συμπεριφορά, διαφορετικέ συμπεριφορέ. Στην πρόσφατη κρίση, η Ισλανδία, μια μικρή χώρα ευρωπαϊκή, επομίστηκε την ευθύνη του τραπεζικού τομέα και πλήρωσε 100% του ΑΕΠ της για την κάλυψη του χρέους. Υπήρξαν άλλες περιπτώσεις όπου αποσύρθηκαν κάποια από το τραπεζικό τομέα, απέσυραν από το τραπεζικό τομέα και έχουμε και μετακίνηση τραπεζών που έφυγαν από τη χώρα του και άνοιξαν θηγατρικέ σε άλλη χώρα, έγιναν πολύ μεγάλες στην άλλη χώρα και όταν αντιμετώπισαν την κρίση απεσύρθησαν. Χρειάζεται θεσμικός, θεσμικό πλαίσιο για να αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα. Ποιο έχει τι ευθύνε, ε, μυθική εταιρεία, θηγατρική κλπ. Χρειάζεται περίπλοκη δομή για να βρει ισορροπία. Είναι η καλύτερη λύση. Εκεί θέλουμε να είμαστε 10-20 χρόνια. Εγώ πιστεύω σε περισσότερη ευρωπαϊκή συνεργασία όμως πιστεύω και σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε δίκαιο συμβιβασμού όπου λαμβάνουμε υπόψη όλα τα συμφέροντα στις ε, αποφάσεις που λαμβάνουμε. Όταν κοιτάμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη θέλουν να κάνουν και άλλες προσπάθειες για την επίτευξη συμβιβασμού. Στα μέσα ενημέρωσης διαφόρων χωρών είδαμε κάποιους να λένε ότι πήγαμε πολύ μακριά, οι αυτοί δεν προχώρησαν αρκετά. Όμως όλοι θεωρούν ότι έκαναν πολλά για να μπορέσουν να πετύχουν τη συμφωνία. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να πετύχουμε κάποια πρόοδο. Εγώ υποστηρίζω περαιτέρω πρόοδο, αλλά θα πρέπει να βασίζεται στην ιδέα σύμφωνα με την οποία μπορούμε να έχουμε διαδικασία λήψεως κοινών αποφάσεων που λαμβάνουν όμως αυτές οι αποφάσει όλα τα συμφέροντα εντό της ενώσεω. Ευχαριστώ. Βίκη. Έχω δύο ερωτήσει. Πρώτο ερώτημα. Το EFMD Κάνατε πολλή δουλειά κι εσείς και οι συνάδελφοι αυτό τον τομέα και προχωρήσατε αρκετά. Αλλά αυτό ξεκίνησε σαν καλή πρόθεση, σαν καλό νομοθέτημα για προστασία του κοινού και του επενδυτή. Αλλά πέρασε βιαστικά το μέτρο. Δεν επληρούσε τι προδιαγραφέ για καλή νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διατύπωση τελική δεν ήταν καλή. Έχει ευρύτερε συνέπειε από ό,τι νομίζαμε αρχικά. Και νομίζω ότι υπήρχαν δύο επιλογές που μπορούσαν να γίνουν εδώ όσον αφορά το θέμα. Είτε συνεχίζουμε σαν Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο να επενδύουμε χρόνο χρησιμοποιώντας τα λαμπρότερα ε, μυαλά που έχουμε στην Επιτροπή μας για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα καλό νομοθέτημα, κάτι που χρειάζεται τεράστιες προσπάθειες και ίσως ε, να μην ανταποκρίνεται στις προθέσεις μας και μπορεί να μας αποσπάσει από άλλες προτεραιότητες που έχουμε και ε, τραπεζικά κεφάλαια, παράγωγα, εποπτεία κλπ. Τα άλλα που αναφέρατε. Είτε, η άλλη επιλογή, ο νέος επίτροπος να πάρει αυτήν την νομοθετική πρόταση, να την επανυποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δει τι υπόθηκε το τελευταίο εξάμεινο, ακολουθεί τους κανόνες περί καλύτερης νομοθεσίας, τις αρχές αυτές και επανέρχεται με μια νέα αφετηρία σε εμά. Ποια από τις δύο επιλογές θα θέλατε να ακολουθήσει ο νέος Επίτροπος. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Το θέμα είναι τι γίνεται. Οι νέες υποπτικές αρχές σε ποιον είναι υπόλογες. Είδαμε τι έγινε τα τελευταία δύο χρόνια. Τεράστια ποσά των φορολογουμένων μπήκαν στα τραπεζικά συστήματα. Έχει απόλυτο δίκιο ο κόσμος. Ζητά σωστό έλεγχο των ρυθμιστικών αρχών. Και όπως γνωρίζετε στο Ηνωμένο Βασίλειο, το FSA είναι υπόλογο στην κυβέρνησή μας και στις εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο φέτος θα πρέπει να διαλέξει το κοινό. Ένα κόμμα θέλει να συνεχίσει το πώς λειτουργεί ο ποπτικός φορέας στο Ηνωμένο Βασίλειο και η άλλη, ο άλλος υποψήφιος θέλει να αλλάξει το σύστημα και να έχει μεγαλύτερο λόγο κεντρική τράπεζα. Χρειάζεται έλεγχος λοιπόν. Αλλά όσον αφορά τη νέα αρχή, οι νέε αρχέ θα διορίζονται, οι επικεφαλεί θα διορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα είναι υπόλογοι αυτοί ούτε στι εθνικέ κυβερνήσει, ούτε στο Κοινοβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο. Άρα έχω ερωτηματικά όσον αφορά τον έλεγχο εκείνων που θα επιφορτήσουμε εμεί με το σύστημα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και θα ήθελα να ακούσω ποιες είναι οι απόψεις σας από αυτό. Άστριντ και μετά πάρα πολύ σύντομα ο Σβέν θέλει να δευτερολογήσει. Ναι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, εγώ θέλω να σταθώ και πάλι στο σημείο αυτό της συζήτησης των λεγόμενων φορολογικών παραδείσων. Υπήρξε μια απόφαση για να εφαρμοστούν τα πρότυπα του ΟΣΑ σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών. Μα υπάρχουν πάντα κάποιοι οι οποίοι κάνουν αυτόματες ανταλλαγές πληροφοριών. Λέτε ότι αυτές οι συμφωνίες δεν επαρκούν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Εγώ πιστεύω ότι η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών δεν οδηγεί σε τίποτα. Γιατί οι φορολογικές αρχές δεν μπορούν <clears throat> να σηκώσουν κεφάλι πάνω από την πλημμυρίδα των πληροφοριών που δεν μπορούν να διαχειριστούν. Πρόσφατα είχε έρθει να με βρει μια κυρία που μου είπε ότι δουλεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά τα έσοδά της είναι στη Γερμανία αλλά φορολογούνται τα εισοδήματά της δεν φορολογούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί δίνονται οι πληροφορίες στις γερμανικές αρχές αλλά δεν φτάνουν οι πληροφορίες σωστά ή δεν τη χάνουν σωστής διαχείρισης και δεν πληρώνει φόρους. Λοιπόν, θα πρέπει επομένω αυτό να αντιμετωπίσετε στην χώρα κατοικία των εργαζομένων. Πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να επανέλθουμε στην πραγματική κατάσταση. Η ίδια η Κομισιόν δέχτηκε να υπάρξει αυτή η αναλλαγή, μάλλον δέχτηκε ότι δεν λειτουργεί η ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά εσείς θέλετε τώρα να καταργήσετε ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί, το οποίο είναι η παρακράτηση στην πηγή, όπως είχε λειτουργήσει αυτή η οδηγία στο παρελθόν. Πρέπει λοιπόν να παραμείνουμε στη γη και όχι να θέλουμε να κάνουμε αυτόματες ανταλλαγές πληροφοριών για τα πάντα <clears throat> και αυτό δεν οδηγεί σε τίποτα λοιπόν. Νομίζω ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μετά από συγκεκριμένη αίτηση είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί πολύ καλύτερα και Πιστεύω ότι η Ισπανική Προεδρία μπορεί να εξασφαλίσει μια συμφωνία προ την κατεύθυνση αυτή. Εγώ δεν καταλαβαίνω δεν αφήνουμε τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν για την, για την φορολογία τη αποταμίευση. Είτε να έχουν ένα σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών, είτε το σύστημα τη παρακράτηση στην πηγή. Τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν την παρακράτηση <clears throat> στην πηγή για τους δικούς τους αυτόχθονες κατοίκους και λειτουργεί μια χαρά. Γιατί λοιπόν να μην γίνει ένα τέτοιο σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τελευταία παρατήρηση, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που αποσύρατε αυτή την πρωτοβουλία που δεν ήταν αρκετά τεκμηριωμένη να αυξήσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα αλκοολικά ποσά. Νομίζω ότι εδώ δεν υπήρχε καν και καμία πρόταση της Κομισιόν για να προχωρήσει κανείς προς την κατεύθυνση αυτή. Ευτυχώς. Κυρία Λούλιν, και εγώ θα ήθελα απλώς να σας πληροφορήσω ότι το άρθρο 11 της τωρινής οδηγίας για την αποταμίευση ζητά από όλα τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών από την στιγμή που πληρούνται οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Αυτό θα γίνει πραγματικότητα σύντομα και επομένω η συζήτηση αυτή μαζί σα θα τελειώσει. Του του τουλεχθέντος υπάρχει και ένα πολύ καλό λόγο για όλα αυτά. Δεν μπορεί κανεί να φορολογήσει το, την περιουσία και τι κληρονομίες χωρί τι απαραίτητε πληροφορίε. Το θέμα θα επιληθεί λοιπόν με την ανταλλαγή πληροφοριών. Σβέν, δεν είναι συζήτηση με την κυρία Λούλινγκ, είναι ερωτήσει προ τον κύριο Υπουργό. Ναι, ήθελα να σας βοηθήσω να καταλάβετε γιατί υπάρχει αυτή η επιμονή εδώ. Εγώ δεν ήμουν ικανοποιημένος με το δικό σας ερώτημα, δική σας απάντηση μάλλον για το, την οδηγία για την αποταμίευση. Πέστε μου και πάλι ποια ήταν τα θέματα που ήταν επίμαχα στο Συμβούλιο και ποια κράτη-μέλη πήρανε θέσεις που οδήγησαν στην εμπλοκή. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ σύντομα κυρία Λούλινγκ, αλλά είναι εκτός μικροφώνου. Εγώ μίλησα για την οδηγία σε ό,τι αφορά την φορολόγηση της αποταμίευσης. Ξέρω ότι προβλέπεται ένα χρονικό διάστημα <clears throat> για την εφαρμογή της. Αν όμως είναι κακή η οδηγία μπορούμε πάντα να επανέλθουμε όταν ξέρουμε ότι δεν λειτουργεί και εξάλλου δεν πρέπει να αναμειγνύουμε την φορολογία των κληρονομιών με τη φορολογία της αποταμίευσης. Yes, um, I Ωραία. Εγώ ξεκινώ με το, την, το ερώτημα που ετέθη σε σχέση με την οδηγία για τους τα εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία. Εδώ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για καλύτερη συνεργασία υπάρχουν θεσμοί οι οποίοι έχουν συστημικά σημαντικό χαρακτήρα που πρέπει να τύχουν ρύθμιση. Δεν είναι αποδεκτό ε, επενδυτικές τράπεζες όπως η Bear Stearns και η Lehman Brothers που ήταν στην, ε, στο κέντρο της κρίσης δεν είχαν την κατάλληλη ρύθμιση. Αν θέλει κάποιος φορέας ο φορολογούμενος να αναλάβει τις απώλειές του και τα προβλήματα στον ισολογισμό του, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα ρυθμιστικό φορέα, μια ρυθμιστική δομή που εξασφαλίζει την εποπτεία των επενδυτικών τραπεζών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ε, ρύθμιση και για τα hedge funds και για τις λεγόμενες εταιρείες private equity, γιατί και οι δύο μορφές αυτές πιστοτικών ιδρυμάτων οδηγούν σε υψηλότερους από το μέσο όρο <clears throat> χρηματοοικονομικούς κινδύνους και επομένως είναι απαραίτητη η ρύθμισή τους όλα αυτά τα οποία περιμένουμε από αυτούς είναι θέματα διαφάνεια. Ότι θα μας εξηγήσουν ποιο είναι το επίπεδο της έκθεσής τους και ποιο είναι το επίπεδο της μόχλεσης, μόχλευσης που χρησιμοποιούνται. Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε καταλογισμό χρηματοοικονομικής ευθύνης χωρίς να ξέρουμε ποια είναι, ποιοι είναι οι κίνδυνοι στην ε, χρηματοοικονομική αγορά. Πρέπει να υπάρξει εδώ μια πρόοδο για αυτά τα θέματα. Δεν είναι να σε μένα να συμβουλεύσω την Κομισιόν τι θα πρέπει να κάνει. Εμεί ακόμα και στι μέρε τη εκπνοή τη Σουηδική Προεδρία θα προσπαθήσουμε να έχουμε πρόοδο. Αλλά υπάρχουν ακόμα μεγάλε διαφορέ απόψε μεταξύ των κρατών Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε σε επίπεδο ΜΕΑ να έχουμε πρόοδο, αλλά αυτό εξαρτάται και από τη στάση των κρατών μελών. Για το θέμα τη ε, λογοδοσία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα γιατί όλοι αυτοί οι φορεί έχουν ενταχθεί σε ένα σαφές σύστημα λογοδοσίας και υπολογότητος μέσα στην ε, Ευρώπη είναι υπόλογα στην Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο. Εγώ δεν θέλω να ξεκινήσω τώρα μια συζήτηση για το ποιοι φορείς θα είναι αυτοί που θα πρέπει να αναλαμβάνουν το ρυθμιστικό έργο. Υπάρχουν πολλά κράτη που είναι έτοιμα να δεχτούν ένα πιο ομοιόμορφο ρυθμιστικό σχήμα όπου θα παίζουν σημαντικό ρόλο οι κεντρικές τράπεζες. Άλλες χώρες όμως δεν θέλουν να έχουν τέτοιου είδους ε, δομές, θέλουν να έχουν δομές όπως τη Βρετανική Financial ε, Supervision Authority. Σε ό,τι αφορά τώρα τις οδηγίες για την αποταμίευση και τους φορολογικούς παραδείσους, εγώ πιστεύω πρέπει να φύγουμε από την, τον φόρο της παρακράτησης και τα θέματα της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Το θέμα δεν είναι μονάχα η συλλογή του φόρου από το εισόδημα των επενδύσεων. Το θέμα είναι να ξέρουμε από ποια επενδυτική δραστηριότητα προήλθε αυτό το εισόδημα. Όσο έχουμε μονάχα φόρο παρακράτησης, δεν έχουμε καμία πληροφορία για την πηγή αυτών των εσόδων και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ε, απόκρυψη των εσόδων ή ακόμα και εγκληματικές ενέργειες, ξέπλυμα χρημάτων κτλ. Πιστεύω θα πρέπει να έχουμε ένα υπεύθυνο σύστημα όπου οι πολίτες πληρώνουν το φόρο τους και τηρείται ο νόμος. Εγώ πιστεύω λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε προς την ε, ε αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που ήταν και στοιχείο της συμφωνίας του 2002. Πρέπει να πω επίσης ότι η δική μου προσδοκία από αυτές τις διαπραγματεύσεις είναι ότι εν καιρό θα επιτύχουμε την πρόοδο θα αποθαρρύνω ίσως Σφεν δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί θα δυσκολεύσω ακόμα περισσότερο τις, ε, αν, τις διαπραγματεύσεις. Οι χώρες που έχουν επιφυλάξεις θα πρέπει να προχωρήσουν και να αλλάξουν την στάση τους γιατί αλλιώς θα έχουμε επανάληψη της διαδικασίας των G20 στο Λονδίνο. Θα έχουμε δηλαδή διεθνείς συμφωνίες που θα είναι προβληματικές για ορισμένες από τις χώρες. Επομένως πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί για να άρουμε τις επιφυλάξεις ορισμένων χωρών. Θα πρέπει να δεχτούν ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή οδηγία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επομένως είναι απαραίτητη η πρόοδος. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να είμαστε πραγματικά ρεαλιστές. Οι χώρες αυτές καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω πρόοδο, ακόμα και εάν δεν, ε, ακόμα και αν υποστηρίζουν ακόμα τις δικές τους θέσεις, κάτι το οποίο θεμητό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Υποθέτω επειδή... Αυτό που απαντήσατε στην κυρία Φόρντ ότι δεν θέλετε να αποσυρθεί η όλη πρόταση γιατί έχετε κάνει τόσο πολλή δουλειά. Κρίμα θα ήταν. Ε, ελπίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε έναν πιο, πιο, πιο καλό συμβιβασμό ε, από αυτόν που είχατε εσείς ε, στο Συμβούλιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά σας.